Good afternoon. Καλησπέρα σας. Good afternoon, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Hey, take your seats in silence. Θύστε σας παρακαλώ. Yes. Good afternoon, everybody. Getting started. Λοιπόν, αρχίζει η συνεδρίαση. Δύο μέρες, σήμερα και αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Αρχίζουμε από την έγκριση της ημερήσιας διάταξη. ακολουθούν ανακοινώσεις του Προέδρου και ήδη έχει έρθει ο πρώτος ομιλητής μας εδώ στο Προεδρείο για να μας ε, μιλήσει για την έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση. Θα ήθελα όμως να αρχίσουμε όσοι ήθεστε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπήρχαν κάποιες αλλαγές, υπήρξαν στο σχέδιο της σημερινής διάταξης ε, και συγκεκριμένα το σημείο 11 το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων. Η συζήτηση ε, δεν θα γίνει στις 45 αύριο, αλλά στις 5.30 το απόγευμα. Διαφωνείτε? Έχουμε σχεδόν όλες τις γλώσσες, εκτός από τα γοδελικά και τα κροατικά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό ε, και εφαρμοστικές ε, πράξεις. Σας έχουν ανακοινωθεί τα σχετικά από το newsletter μας. Εσωτερική προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων έχει οριστεί και σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Γι' αυτό παρακαλείστε να έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες σας και να το διαδώσετε ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 11, 11.30. Ε, ας αρχίσουμε όμως ε, τώρα με το θέμα ουσία το πρώτο. Έκθεση πρόοδου σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση. Θα ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση που καλωσορίζουμε και τον ομιλητή μας, τον κύριο ε, Μίχελ Μάικαλ Σότερ, Διευθυντή για τη Μετανάστευση και την Προστασία στη Γενική Διεύθυνση Home Εσωτερικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσκαλέσαμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει την έκθεση πρόοδου της σχετικά. Αυτό γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βλέπουμε ποια είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που ε, αποφασίστηκε αυτό το 2015. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη παρουσίαση γιατί είναι η τελευταία πριν αναλάβει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεση καταλήγει με μια παρατήρηση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Αλίμονο. Ε, το ευρωπαϊκό σύστημα, το κοινό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου θα πρέπει να απεμπλακεί επιτέλους στο Συμβούλιο, να ενισχυθεί για να τεθεί σε ισχύ και να μπορούμε να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται ε, την προστασία μας. Και θα πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμες οδούς να φτάνουν εδώ ε, όσοι ζητούν άσυλο και όσοι αναζητούν εργασία και μεταξύ αυτών επίσης εργασίες υψηλών προσόντων. Γιατί ακόμα αυτοί οι διάβλοι δεν υπάρχουν νόμιμοι. Για το λόγο αυτό περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίαση και θα γίνει και συζήτηση. Έχει προγραμματιστεί μία ώρα για τη συζήτηση αυτή και προτείνω να πάρει το λόγο ο κύριος Σότερ για 10 λεπτά για να μας μείνει χρόνος και για τη συζήτηση για τα μέλη μας που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και να ακούσουν και τις απαντήσεις. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε να παρουσιάσω την έκθεση πρόοδου του Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μετανάστευση. Όπως αναφέρατε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Εξετάζουμε τα βασικά επιτεύγματα όσον αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο που επετεύχθη μετά το 2015 εστιαζόμενοι ιδιαίτερως επί των αναλυφθέντων βημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την έκθεση προόδρου του Μαρτίου 2019. Αν επιτρέπετε να ξεκινήσω παρουσιάζοντας την κατάσταση όσον αφορά τις διάφορες διαδρομές μετανάστευσης. Καταρχάς, γενική εικόνα. Η έκδοση παρατηρεί ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα πρώτης κρίσεως. 19. το 2019 μέχρι τέλος Οκτωβρίου ήταν περίπου 92% χαμηλότερες από ότι την ίδια περίοδο του 2015. Πιο συγκεκριμένα, Ανατολική και Δυτική Μεσόγειος. Σημαντική αύξηση είδαμε στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως προς Ελλάδα και Κύπρο και στα Δυτικά Βαλκάνια αναλόγως με περίπου 7.400 αφήξεις το 2019 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Οι αφήξεις από την άλλη στις δυτικές ακτές της Μεσογείου μειώθηκαν σημαντικά το 2019. Περίπου 27.300 αφήξεις μέχρι 3 Νοεμβρίου. Στο δυτικό άκρο της Μεσογείου βλέπουμε μείωση 50% εν συγκρίση με την ίδια περίοδο πέρσι. Την περασμένη εβδομάδα ο γενικός μου διευθυντής ήταν εδώ και σας μίλησε για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα έχει υποστεί πολύ έντονες μεταναστευτικέ πιέσει επί σειρά ετών. Όμως, όπως γνωρίζουμε, τα προβλήματα που εντοπίζει η Ελλάδα στη διαχείριση της μετανάστευσης δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, είναι θέμα ευρωπαϊκό επίσης και απαιτείται μια απάντηση ευρωπαϊκή. Κατεπίγουσες δράσεις αποφασιστικής σημασίας χρειάζονται για να ανακουφιστεί πίεση στα νησιά και να βελτιωθεί η κατάσταση για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Κυρίως να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών και θα πρέπει οι δυνατότητες υποδοχής εκεί να αυξηθούν και στην υπηρετική χώρα. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση κυρίω εν ώψη του επικείμενου χειμώνα. Αποτελεσματικότερες διδικασίε ασύλου θα συμβάλλουν τα μάλλα στη βελτίωση της εξεργασίας των ετοιμάτων ασύλου και έτσι να επιταχυνθεί η επιστροφή εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα διαμονή και παραμονή. Σχετικά με αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε τη διαδικασία θέτηση τη νέα ελληνική νομοθεσία για την υποδοχή και το άσυλο. Εκ του σύνεγγυ γνωρίζουμε ότι η νομοθεσία υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στι 31 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα την 1η Νοεμβρίου. Και ενώ περιμένουμε την πλήρη κοινοποίηση και ενημέρωση τη νομοθεσία για να αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν συμμορφούνται ο νόμο με το νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ήδη οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησαν ανάλυση του κειμένου που έχουν στα χέρια του, ούτω ώστε να εξασφαλίσουν ότι συμμορφούνται πλήρω με το κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Βεβαίω, ευπρόσδεκτοι στόχοι που έχουν τεθεί για το νέο νομοσχέδιο δηλαδή επιτάχυνση και αποτελεσματικότητες διαδικασίες. Θέλουμε όμως να δούμε ότι ποτέ δεν θα υπάρξει καμία υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας αυτών. Για την Κεντρική Μεσόγειο, στρέφομαι στην Κεντρική Μεσόγειο, τι βλέπουμε εκεί, ότι παρά σημαντική αύξηση αφήξεων προς Μάλτα, με περίπου 3.100 μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, δηλαδή 200% αύξηση σε σύγκριση με την περσινή ανάλογο περίοδο. Γενικά, οι αφήξει στην κεντρική Μεσόγειο παρατύπω μεταναστών παραμένουν μικρές, 13.000 αφήξει για την ίδια περίοδο. Αυτό είναι 44% μείωση εν συγκρίση με την ίδια περίοδο πέρσι. Αυτή η κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο πόρο απέχει από την πρώτερη εμπειρία περίοδο 2015-2017. Τώρα, άλλο να μιλάμε για φίξεις και άλλο να μιλάμε για την πίεση επί του συστήματος ασύλου όσον αφορά τις αιτήσει του ασύλου, τι βλέπουμε όσον αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταθεροποίηση όσον αφορά την πίεση επί των εθνικών συστημάτων ασύλου μέσω όρο αιτήσεων που είναι χαμηλότερο σημαντικά το 2019 σύγκριση με την ακμή το 2015 με 2016, αλλά ο μέσος όρος είναι ακόμα υψηλότερος από ό,τι πριν από την κρίση. Αυτά όσον αφορά τις αιτήσει ασύλου. Όσον αφορά τις παράνομες διελεύσεις συνόρων, τις παράτυπες διελεύσεις συνόρων, είδαμε ότι οι παράτυπες αυτές διελεύσεις το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31 Οκτωβρίου ήταν 103.000 περίπου, χαμηλότερο στοιχείο που έχουμε αριθμητικό στοιχείο την τελευταία πεντέτια, αυτή την περίοδο τη χρονική του έτους. Τώρα, στρεφόμενος προς τα γενικά επιτεύγματα, μπορούμε να πούμε ότι εν γέννη η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια συλλογικά κατάφερε να θεσπίσει μέτρα για τη δημιουργία ενός ολιστικού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ξαναδημιουργήσαμε κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για παγίωση των μέτρων και βελτίωση και διεύρυνση του νομικού μας πλαισίου και των επιχειρησιακών μέτρων. Παρ' όλα αυτά, εν γέννη, είναι ισχυρότερη η διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει αλληλεγγύη παρέχεται υποστήριξη στα κράτη-μέλη Ένα τμήμα του γενικού πλαισίου που ανέφερα συνεπάγεται συνεργασία με τρίτε χώρε. Έχουμε τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, Τουρκία, Φερρυπίν, εν είδη παραδείγματο. Την περασμένη εβδομάδα η Γενική Διευθύντριά μου συζήτησε το θέμα αυτό μαζί σα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η δήλωση είναι σημαντικότατη και θα συνεχίσει τι προσπάθειε να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή αυτή. Αυτό απαιτεί προσπάθειε ε, πανταχώθεν. Αναφερόμενος στη δυνατότητα φιλοξενίας προσφύγων στην Τουρκία, εκεί βλέπουμε ότι παρέχεται υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 97% των 6 δις ευρώ των πόρων για το μέσο διευκόλυνσης έχουν διατεθεί και οι εκταμιεύσεις μέχρι τώρα είναι περίπου 3 δις. Αυτό το μέσο για τη διευκόλυνση μετανάστευση παρέχει υποστήριξη για καθημερινέ ανάγκε για τα παιδιά που στο σχολείο, για υγεία, εκπαίδευση σε γλώσσε κλπ. Αυτό το μέσο έδωσε τη δυνατότητα για εμβολιασμού, ε, πρόνοια, πρόσβαση σε γιατρού και κέντρα υγεία για του μετανάστε. Ε, γενικότερα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. όλο ιδιαίτερο θέλω να αναφερθώ στην υποστήριξη την οικονομική υπόδοση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Πάνω από 2,2 δις ευρώ για υποστήριξη από το 2015 και μόλις πρόσφατα, το Σεπτέμβριο του 2019, άλλα 8 εκατομμύρια διετέθησαν μέσω ε, δύο δόσεων κατεπίγουσας ε, βοήθειας στη Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για να ανοίξουν κέντρα στέγασης στην Υπηρετική Ελλάδα και για τη διαφύλαξη ε, των παιδιών που διέρχονται τα σύνορα σε σημεία διέλευσης δεν έχουν επιτευχθεί τα πάντα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα σύλλου και την εφαρμογή αυτού. Δεν έχουμε κατορθώσει να συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί του νομοθετικού πλαισίου. Σημειώθηκε πρόοδος. Σε πέντε από τις προτάσεις το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο ευκταίο αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρήσετε ότι άοκνα θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει κοινό τόπο, ώστε να προχωρήσουμε προς δίκαια αποτελεσματικότερη βιώσιμη προσέγγιση του ασύλου και να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα για ασύλου. Σημειώθηκε πρόοδος για νόμιμες διόδους για εκείνους οι οποίοι χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί σαν μία από τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελευταία χρόνια κυρίως από ό,τι φαίνεται από τους αριθμούς εκείνων που έχουμε αντικατασταθεί, ε, πάνω από 63.000 άτομα έχουμε αντικατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 και βλέποντας τα γίνει στο μέλλον, συνεχίζεται η προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απίθυνε έκκληση για συνέχιση της μετακατάστασης το 2020. Κάτι μέλη επιβέβαιωσαν την υποχρέωσή του να δώσουν δυνατότητα αντικατάσταση στο μέλλον και είδαμε δεσμεύσεις για άλλες 30.000 θέσεις. Και τώρα Βλέπουμε τι θα γίνει με τη σχετική χρηματοδότηση για να επιτευχθεί αυτό. Τώρα να στραφώ προς το θέμα των επιστροφών και πανισδοχών. Καταλαβαίνω ότι χρονοτριβώ κάπω, ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Όταν μιλάμε για πλήρη πολιτική, υπάρχουν πολλά σημεία να καλυφθούν όσον αφορά τι επιστροφέ και πανισδοχέ. Οι πρόσφατε συμφωνίε και διευθυντή επανεισδοχή έχουν συναυθεί με 23 χώρε προέλευση και διέλευση, με πρόσθετη υποστήριξη για αποτελεσματική επιστροφή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η έκθεση όμω διαπιστώνει ότι χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια προ βελτίωση των γενικών αποτελεσμάτων στο μέλλον. Λοιπόν, προσβλέπουμε στον κώδικα για τι θεωρήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που δίνει τη δυνατότητα κατά περίπτωση καθορισμού τη προσεγγίσεω μαζί με τι χώρε εταίρου υπό το φω τη συνεργασία που επιτυγχάνεται στην επανεισδοχή. Αυτό είναι κάτι που θα τεθεί σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2020. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μέλλον. Συνεχίζουμε την εφαρμογή μέτρων στο βάση του σχεδίου δράσεω για την παράνομη διακίνηση των μεταναστών για να εμποδίσουμε τις εγκληματικέ οργανώσεις να κινούνται σε αυτό το τομέα. Και έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Το αναφέρει η έκθεση στον Ήγηνα μέσω κοινή ομάδα έρευνα που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του καταπιστεύματο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μετά, δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη ε, λαθροδιακίνηση μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διενεργεί έρευνε και θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινέ επιχειρησιακές συνεργασίες με χώρες εταίρου. Ένα από τα μέτρα που εθέτησε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2018. Τώρα για τα εξωτερικά σύνορα και το έργο τη Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Μαθηροφυλακή και του σχετικού οργανισμού συνεχίζεται η προσπάθεια να ακολουθούμε διαχείριση συνόρων ολοκληρωμένη μέσω της εφαρμογής του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και την Μαθηριακή Έλεγχο των Συνόρων. Η δεύτερη φάση ενίσχυσης λοιπόν του, ελέγχου των συνόρων και των ακτών τι συνεπάγεται ότι ακτοφυλακές των κρατών μελών και η υπηρεσία ακτοφυλακής ε, κινούνται από κοινού. Αυτή είναι η εφαρμογή του κανονισμού του 2016. Βέβαια, χάρη και στι προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα επιτυχαίνουμε όλα αυτά και είχαμε και μεταρρύθμιση του υποκείμενου κανονισμού για περαιτέρω ενίσχυση τη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του οργανισμού φύλαξων συνόρων με 10.000 προσωπικό και περισσότερο επιχειρησιακό εξοπλισμό κοινό που θα διαχειρίζεται ο οργανισμό αυτό φύλαξη των συνόρων από τη στιγμή που τελικά θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμό, νομίζω το Δεκέμβριο, θέλουμε να μπούμε στη δεύτερη μεταρρύθμιση του οργανισμού για τα σύνορα, κάτι που υποστηρίζεται από δικό χάρτη. Πολλά πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε τα 10.000 μέλη του προσωπικού να μπουν στις σωστές θέσεις. Στρεφόμενο στη Λιβύη τώρα, ξέρω ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει πολύ ανησυχητική. Πρέπει να επιταχύνουμε την εκένωση των πλέον ευαλώτων ατόμων, να αυξηθεί η επιστροφή και ο ρυθμός μετεγκατάστασης στα πλαίσια του ε, κατεπήγοντος μηχανισμού μετακίνησης. Μετά από την εκένωση που ξεκίνησε το 2017 στη Λιβύη και μέχρι 5 Νοεμβρίου, Συνολικά 4.024 άτομα συμπεριλαμβανομένων συνοδεύτων ανηλίκων έχουν εκενωθεί. Τώρα, αν επιτρέπετε να ολοκληρώσω κάπως, να κλείσω, κάναμε πραγματική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιούργησαν νέα προβλήματα και προκλήσεις αναφέρομαι προς προσφατά στην κατάσταση στη Βόρεια Συρία. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τα μέσα προβλήματα και να συνεχιστούν οι δρομολογηθήσεις εργασίες θα πρέπει όλος ιδιαίτερος να επιμείνουμε ε, όσον αφορά τις αυξήσεις της αυξημένης Ανατολική Μεσόγειο να εξασφαλίσουμε βελτίωση των συνθήκων στα νησιά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θα εξακολουθεί να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα παρόλο που η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία. Βέβαια, πρέπει να παρακολουθούμε του σύνεγγυ τις ζωές που έχουν διασωθεί στη θάλασσα, να συνεχίσει την προσπάθεια η διάσωση ζωής στη θάλασσα, να υπάρχουν οι σωστές λύσεις για την υποβίβαση αυτών των ανθρώπων. Τον τελευταίο χρόνο είδαμε ad hoc λύσεις μετεγκατάστασης που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα όμως. Κινηθήκαμε προς κάπως πιο προβλέψιμο πλαίσιο, ευπρόσδεκτο αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό το φως της κοινή δηλώσεως προθέσεων που συνήθει από Μάλτα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία στις 23 Σεπτεμβρίου. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος ευρωπαϊκού για το άσυλο. Σταματάω εδώ και με τα χαράς να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε στις 5 θα έρθει ο Επίτροπος Τζούλιαν Κίνγκ για να μιλήσει για την ατζέντα του. Ε, λοιπόν, μια μισή ώρα να ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη και μετά ε, εσείς θα απαντήσετε. Για το ΕΛΚ η κυρία Ντουπον Ναι, επειδή δεν βλέπω συντονιστή του ΕΛΚ θα σας δώσω λόγο σε εσά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συντονιστές. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σόρτα για την παρουσίασή σας. Νομίζω μας έδειξε ξεκάθαρα πόσο περίπλοκο και δύσκολο είναι το θέμα, αλλά και μια συνολική στρατηγική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ταυτόχρονα ότι χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική. Μιλήσατε και για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που δεν έχουν μειωθεί γύρω μας. Ε, δείχνουν οι ε, πρόσπατες εξελίξεις ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια κοινή στρατηγική. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα επιμέρους θέμα που αναφέρετε και εσείς που είναι εταιρική σχέση με τρίτες χώρες για τις επανεισδοχές και επιστροφές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 23 χώρες με τις οποίες έχουμε διαπραγματευτεί συμφωνίες και ε, καλές συμφωνίες σε μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα ο αριθμός όμως των ενδιαφερομένων είναι σχετικά μικρός για επιστροφές και επαναπροωθήσεις. Ε, οι επανεισδοχές καλύτερα. Ε, ποιες είναι οι δυνατότητες που βλέπετε εκεί, ε, τι μπορείτε να προτείνετε για να καταπολεμηθεί ε, το οργανωμένο έγκλημα, να δημιουργηθούν νόμοι μεσοδοί, αλλά ενδεχομένως και νέες μορφές οικονομικής συνεργασίας, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα με μονομένων κρατών μελών που βοηθούν ε, και για τη μετανάστευση και προωθούν και την οικονομική ανάπτυξη στις δικές μας κοινωνίες. Ε, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση, γιατί κύριε Σότερ, εσείς μιλήσατε για κρίση. Η κρίση δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται σε εμά, αλλά με το γεγονός μάλλον ότι τα κράτη-μέλη μας δεν είναι σε θέση να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Ισχυρίζομαι ότι και το τρέχον σύστημα ασύλου που, δεν, ε, που ισχύει εδώ και καιρό δεν εφαρμόζεται παντού. Η καταγραφή ε, των προσφύγων που φτάνουν δεν διεκπεραιώνεται γρήγορα και διαιωνίζονται οι ε, διαδικασίες ασύλου. Σε πολλές χώρες είναι τρομακτικές οι διάρκειες και πολλές φορές δυσκολεύουν τη ζωή των προσφύγων έτσι να ενταχθούν γιατί δεν ξέρουν αν θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, αν θα πάρουν άσυλο και αν θα παραμείνουν. Όλα αυτά δυσκολεύουν και τη ζωή των δικών μας πολιτών επιτόπου. Έχω να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους αριθμούς. Μιλάτε για 150.000 παράτυπους μετανάστες πρόσφυγες που έφτασαν το 2018 στην Ένωση. Μα η Ήπειρο μα έχει 500 εκατομμύρια κατοίκου Κανονικά αυτό δεν θα έπρεπε να ήταν πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε είναι με την επανεκατάσταση, το relocation. 34.700 είναι το σύνολο των όσων έχουν κατανεμηθεί και επιμεριστεί. Μα τι γίνεται με τους υπολείπους. Οι περισσότεροι παραμένουν στις χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα. Και όλα τα υπόλοιπα κράτη, όλα τα υπόλοιπα κράτη ε, είναι τελείως αλληλέγγυα στη συμπεριφορά τους. Θα μπορούσατε να μας πείτε εάν μπορεί να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Δεύτερον, και στην επανεκατάσταση, αλλά και στη μετεγκατάσταση, το resettlement, Όλα αυτά που μας λέτε είναι γεγονότα ή είναι υποσχέσεις των κρατών μελών. Γιατί αυτά είναι ωραία και πιασάρικα στον τύπο, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Ε, και μετά τι γίνεται με τους πρόσφυγες που έχουμε φέρει από τη Λιβύη μέχρι τώρα που έχουμε εκενωθεί. Εμείς ακούσαμε για 49.000 σύνολο. Έχει στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που παραμένουν ακόμα σε αυτή την παγίδα της Λιβύης. Η κυρία Νετβέλτ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και η κυρία Ζίπελ, θα ήθελα να αναφερθώ στην φρασιολογία που χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε για κρίση, για τη μη δυνατότητα ή την μη βούληση για να βρεθεί συμφωνία από του 28 από τα 28 κράτη-μέλη. Ε, κατεφημισμό λέμε κρίση βέβαια. 28 ηγέτε από υποτίθεται πολιτισμένα κράτη-μέλη τη Ένωση δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ του, αλλά πολύ εύκολα βρίσκουν συμφωνίε με τον κύριο Ερντογάν. Με τον κύριο Ασάντ τώρα. Κάποια κράτη-μέλη φτάνουν ε, ε, κοντά στο Χασάπι Ασάντ. Με ένα στόχο και μόνο να στείλουν ανθρώπους πίσω στη Συρία υπάρχουν και βρώμικες συμφωνίες μεταξύ κάποιων κρατών μελών και τη Λιβύη και αυτό είναι ντροπή. Η συνάδελφος από το ΕΛΚΑ αναφέρθηκε πριν ε, την συνεργασία, για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση, τη σύμπραξη. Δεν είναι συμπράξεις αυτέ. Είναι βρώμικες συμφωνίε για να φτιάξουμε ένα οχυρό που λέγεται Ευρώπη. Να μιλάμε καθαρά. Έχω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα να θέσω για τη συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει σημαντική μείωση παράτυπων ε, αφήξεων. Πολλά χρήματα έχουν δοθεί στο Μαρόκο, ε, περίπου 250 ε, εκατομμύρια. Ε, λέει η Κομισιόν όλα πάνε καλά, ε, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Εγώ έχω ερωτηματικά. Πρόσφατα είχαμε μια υπόθεση ενός Ολλανδού υπηκόου, μαροκινής καταγωγής, που, που επέστρεφε από τις διακοπές του και στα σύνορα του πήραν το διαβατήριο χωρίς καμία εξήγηση, τον άφησαν στο δρόμο, δεν είχε κανένα να τον ε, ε, εκπροσωπήσει και δεν του είπαν καν γιατί του πήραν το διαβατήριο. Αυτή είναι η νέα πολιτική, αυτή είναι η νέα διαχείριση της μετανάστευσης. Για την Τουρκία τώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη δήλωση συνεργασίας με την Τουρκία λέει, λέτε ότι οι συζητήσει μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζονται για να υπάρξει ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερη συνεργασία στη διαχείριση τη μετανάστευση. Τώρα μιλάμε για διαχείριση τη μετανάστευση, ε, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για τη σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, ε, και αυτό κατά φημισμό το λέμε. Ε, μπορείτε να μα εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι συμβαίνει με βάση τη νέα κατάσταση. Επίση, επανεκατάσταση από τον Ήγυρα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο ενθουσιώδη τα κρατη να λαμβάνουν, να δέχονται μετανάστες μετά από κατάσταση παρότι έχουν συμφωνήσει. Έτσι λοιπόν ε, εδώ διακυβεύεται η εκένωση της Λιβύης, ε, εκένωση από τη Λιβύη. Επίσης αναφέρεται σε πιλωτικά προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση, αλλά πολύ λίγα πράγματα και λίγος ενθουσιασμός κυρίως ε, υπάρχει σε πρωτοκρατό μελών. Πώ θα λειτουργήσει αυτό ή πώ δεν λειτουργεί αυτό, ποια κράτη-μέλη συνεργάζονται, ποια όχι και τι θα κάνουμε για να συνεργαστούν. Ευχαριστώ κυρία Τρίκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάτε για την παρουσίασή του. Ε, που μας αναφέρθηκε και το τι γίνεται στην, σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντα την έκθεση είναι ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον αριθμό των παράτυπων αφήξεων. Και το συμπέρασμα είναι ότι έχει μειωθεί ε, σε ό,τι αφορά πολλές οδούς αλλά αυτή η μείωση σχετίζεται με την αύξηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Μεταξύ αυτών των παράτυπων μεταναστών υπάρχουν και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι ζητούν προστασία, ζητούν πρόσβαση σε μια διαδικασία ε, χορήγησης ασύλου. Όταν διαβάζουμε έκθεσης, ε, εκθέσεις για τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ε, στην Κροατία, παραδείγματος χάρη, όπου πρόσφατα αποφασίσαμε ότι συμμορφώνονται επαρκώς για να ε, ενσωματωθούν στη Σέγγεν. Η Ισπανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία. Εκεί ε, ακούμε συχνά για αποθήσεις, για pushback. Ε, πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε τα, τα πρότυπα που έχουμε θέσει. Τι κάνει η Κομισιόν, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου αλλά και για τα τι άλλε προδιαγραφέ που στα πλαίσια του, ασύλ, του, του, του κεκτημένου για το άσυλο. Επίση ε, υπάρχουν και οι χώρε transit. Πολλοί, πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Τι θα γίνει με τα συστήματα ασύλου εκεί. Ε, επίσης, επειδή μιλάμε για αλληλεγγύη, ο αριθμό ε, ε, των ε, επανεισδοχών έχει αυξηθεί, ωραία, αλλά ποιο είναι η ακριβή φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και να αφήνουμε την Τουρκία και άλλες χώρες ε, να κάνουν τη δουλειά για μας. Ποια είναι η φιλοδοξία μας και τι θα ήταν αναλογικό για μας σε σχέση με αυτά που ζητάμε για τρίτες χώρες τώρα και τέτοια τη relocation τώρα. Ε, είδαμε τα στοιχεία την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία ε, που ζητούν μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή προσέγγιση αλληλεγγύης όχι μόνο αυτά τη δήλωση τη Μάλτα. Ε, Εσεί λέτε ότι πρέπει να έχουμε μια δομημένη προσέγγιση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μπορεί να πάρει χρόνο, όσο ε, χρόνια όσο το, το κάνουμε αυτό. Τι θα κάνει η Κομισιόν στο, μεταξύ για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αλληλεγγύη. Ο κύριο Ταρντίνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Διάβασα την έκθεση. Βρήκα τα αναμενόμενα. Βλέπουμε ότι κάναμε μεγάλη πρόοδο, ότι ήμασταν πολύ καλοί, μεγάλη πρόοδο που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά γνωρίζουμε προφανώς δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Και έγινε παραδεκτό και στην ίδια την έκθεση αυτό παραθέτει αυτό λεξί, αυτό που λέτε, ότι όλες οι πτυχές αυτής της δουλειάς έχουν κλωθεί. αντίθετα λέτε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση ενός νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πλήρω και βιώσιμο πλαίσιο όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο. Πότε λοιπόν θα συμβεί αυτό. Διότι αυτό μας το είχατε πει, μας το είπε και η Επίτροπος στην Ακρόαση. Το είπε και ο, ο κύριος ε, Αβραμόπουλος εδώ και πέντε χρόνια. Και όλη την πενταετία αυτό λέτε. Ενώ βλέπουμε χιλιάδε αποβιβάσει, ε, εκατοντάδε ε, θανάτου στη θάλασσα, δεν άλλαξε τίποτα. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Βαντελάιν, μιλάει για ένα κοινό σύμφωνο για τα άσυλο και μετανάστευση. Κατά λοιπά, πρέπει να αρκεστούμε σε μια συμφωνία, τη συμφωνία τη Μάλτα, που η Ιωνή έγινε αστεία εκεί, βλέποντα πώ εφαρμόζεται στην πράξη. Μετά λέτε ότι είναι θεμελιώδη εταίρο μα η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ε, θα με 6 δισεκατομμύρια ευρώ την κυβέρνηση ε, Ερντογάν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Είναι χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου και υπάρχουν απειλέ από την Τουρκία για νέε ροέ προ την Ευρώπη και λόγω γενική κατασταση. Τι πρέπει να κάνετε, πώ θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σήμερα δείχνουν την καθιστική ατάξα. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο μέλλον. Η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματο, του κοινού συστήματο ασύλου πρέπει να επιλύσει όλα τα προβλήματα, ακόμα ε, Λοιπόν, έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ε, δεν υπάρχει κατάλληλη συμμετοχή στο σύστημα. Χρειάζεται αλλαγή προσέγγισης. Λοιπόν, αυτό το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται μια παρουσία στην αφρικανική επικράτεια, ούτω ώστε να δημιουργηθούν εκεί πραγματικά hot spots και να μπορούν, ε, ε, να μπορούν ε, εκεί πέρα να ελέγχονται άνθρωποι που θέλουν να έχουν τις ευρωπαϊκές ακτές. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε τελικά όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιο εκπρόσωπο του ECR. Θέλετε εσείς Παρακαλώ, κυρία Κενκό. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Δεν έχει σημειωθεί πρόοδο ε, αυτό το διάστημα. Η Κομισιόν ε, θα επικεντρωθεί στην σωστή εφαρμογή τη υπάρχουσα νομοθεσία και πώς ο κανονισμός του Δουβλίνου λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ξεκίνημα της ε, μεταστευτικής κρίσης. Κυρία Μπιόρκ για την ΚΟΕ, ναι, ευχαριστώ. Πρέπει να πω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ε, σοσιαλδημοκράτες, αλλά και από την ομάδα Renew, ότι πιστεύω ότι πραγματικά εδώ μας λείπει λίγο μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Αν σκεφτούμε πώς, ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με τη σύμβαση τη Γενέβη, τι κάνουμε σε ό,τι αφορά ζωέ στη τη θάλασσα, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, το κράτος δικαίου. Εάν έχει δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη με βρώμικες συμφωνίες ε, πολιτοφυλακές της Λιβύης ή με τον Ερντογάν στην Τουρκία, κάποιοι κοιτάζουν και προς το χασάπια σάδια συμφωνίες πλέον, δεν πρόκειται για αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ε, εν δεν θέλουμε να οικοδομήσουμε τέτοιου εμπιστοσύνη. Θα ήθελα αντιθέτω, πέρα από του αριθμού που μειώνονται των αφήξεων, θέλω να μα πείτε πόσου τελικά προστατεύσαμε. Το λέει η έκθεση, αλλά πόσου προστατεύουμε. Ε, τι πετυχαίνουμε σε σχέση με άλλε χώρε, με άλλε υπήρου, που επίση δίνουν προστασία σε ανθρώπου που τη ζητούν. Σε σχέση με αυτού, ποια είναι η δική μα θέση και τι γίνεται με τη διάσωση στη θάλασσα. Τι κάνουμε για να μην ποινικοποιούμε αυτού που βοηθούν του πρόσφυγε και τι θα κάνουμε για να σταματήσει η συνεργασία με τις πολιτοφυλακές της Λιβύης. Ε, εδώ θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει στο δικαστήριο για κρίματα κατά της ανθρωπότητας και για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις ε, και πολλά στοιχεία που μιλούν για απόθυση ε, που γίνονται στο όνομα της Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλους, ε, με χρηματοδότηση δική μα δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα. Ιδάλω θα μπλέξουμε και κάτι ακόμα. Εξηγήστε μας ε, πώς μπορούμε να μιλάμε για επιτεύγματα, ε, πώς μπορούμε να έχουμε κάποια, ε, κάποιες προδιαγραφές αξιοπρέπειας Το Δεκέμβριο στη Γενέβη θα λάβει χώρα το Φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΗΠΑ. Έχουμε πάρει θέση για την ε, επανεγκατάσταση ότι πρέπει να είναι ένα εργαλείο ε, προστασία. Δεν πρέπει να συνοδεύεται από προποθέσει. Ε. Δυστυχώ το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται ω εργαλείο για συμφωνίε για παζάρια με τρίτε χώρε, ενώ δεν, έχει δημιουργηθεί για κάτι τέτοιο. Δεν, δεν έχει δημιουργηθεί για αυτό το λόγο. Τι θα γίνει λοιπόν με τους αριθμούς. Οι αριθμοί δεν είναι αρκετά υψηλοί, δεν υπάρχει μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση. Αναμένουμε περισσότερε δεσμεύσει ε, το Δεκέμβριο εκεί στη Γενέβη. Ο κύριος Τομπέ έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, να ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσίαση. Ε, οι περισσότεροι από εμά ε, μακροπρόθεσμα Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Για μένα είναι σαφές ότι είμαστε μακριά από, την, από το να φτάσουμε στην πρόοδο. Δεν υπάρχει κοινή θέση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σαφές πολιτικά μεταξύ κρατών μελών αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα είναι σαφές ότι ένας τρόπος να προχωρήσουμε είναι να έχουμε ένα πιο σαφή διαχωρισμό μεταξύ των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων. Και θα ήταν καλό ο Διευθυντής να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Πώς το βλέπετε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές για να γίνει πιο σαφής ο διαχωρισμός αυτός. Ευχαριστώ η κυρία Μπούρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, κατάλαβα Μπουρχαρτ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Σπούρεκ. Υπάρχει το θέμα των ε, μεταναστών για κλιματολογικού λόγου. Φεύγουν από τι χώρε του λόγω τη κλιματική αλλαγή. Και ο αριθμό των ανθρώπων αυτών θα αυξάνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ω τώρα δεν έχει αναγνωρίσει κλιματικού πρόσφυγε η σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες δεν τους καλύπτει επίσης. Η σύμβαση αυτή έχει εργαστεί, έχει προσπαθήσει να δει ποιε θα είναι οι επιπτώσεις, οι πολιτικές ε, της αυξανόμενης μετανάστευσης για κλιματικούς λόγους. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλσαλάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία ε, κύριε για την παρουσίαση. Εγώ όταν ασχολούμαι με θέματα μετανάστευση είναι δύσκολο να δω το θέμα των ροών των μεταναστευτικών ως κρίση. Διότι και εγώ ήμουν μετανάστρια για 15 χρόνια. Και είναι μια προσωπική καταστροφή. Ε, αυτή είναι η δική μου προοπτική. Αν μιλάμε λοιπόν για καταστροφή και για κρίση, αυτή ισχύει για του πρόσφυγε, όχι για την Ευρώπη. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπαν και κάποιοι συνάδελφοι πριν από μένα. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Στην έκθεσή σας λέτε ότι η παράτυπη ε, των συνόρων αυξάνεται στα Δυτικά Βαλκάνια. Και την περσμένη εβδομάδα συνάντησα κάποιε ε, ΜΚΟ από τη Βοσνία που ανησυχούν για το πώ η κυβέρνηση προσεγγίζει την κατάσταση αυτή με τους μετανάστες και πώς ε, αυτοί οι μετανάστες ή και οι πρόσφυγες ζουν υπό άθλιες συνθήκες χωρίς καμία αξιοπρέπεια. Ε, δίνουμε χρήματα στους Βόσνιους αλλά δεν παρακολουθούμε τι γίνεται μετά με τα χρήματα αυτά και πολλές ΜΚΟ ε, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση αυτών των εργασιών. Ποια είναι η άποψή σα, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε εμεί ω ε, θεσμικά, θεσμικά όργανα τη Ένωση την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων όταν τι ξεμαρτωτούμε εμεί. Η κυρία Μπουρκχαρτ. Θα μιλήσω στα γερμανικά, λέει ο κύριος Μπουρκχαρτ. Ε, για το θέμα της Κροατίας να συνεχίσω κι εγώ. Με ενδιαφέρει, γιατί δεν το διάβασα στην έκθεση. Υπάρχουν ε, ε σε γνώση σας στοιχεία για τα pushback, για τις αποθήσεις. Ε, πρώτη ερώτηση, τα ξέρει αυτά η Ευρώπη. Δεύτερη ερώτηση, στη σελίδα 5 ε, λέει η έκθεσή σας ότι 100.000 Αφγανούς λέει θέλετε να τους στείλετε πίσω στην Τουρκία. Δεν λέει εκεί όμως ότι εξήγηλε ο κύριος Ερντοάν ότι θα στείλει ε, ξανά στη Συρία 2 εκατομμύρια Σύρους. Αυτό σας έχει διαφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι στάση έχετε. Γιατί έτσι δεν θα μπορούμε να στέλνουμε σύρους στην Τουρκία, γιατί θα υπάρχει αλυσιδωτή απέλαση. Το τρίτο, πολύ καλά, ε, ε, ε, το θεωρώ θετικό αυτό, ότι θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Τι θα γίνει φέτος διαφορετικό, γιατί τέσσερα χρόνια εδώ συγκρίνουμε την κατάσταση με τα ελληνικά νησιά και κάθε χρόνο έχουμε τις ίδιες αιτήσει και αιτήματα και δεν αλλάζει τίποτα. Ε, ο Υπουργό Ζεχόφερ Εσωτερικών τη Γερμανία πρότεινε ένα νέο σύστημα ασύλου. Το Μάρτιο, λέει, Απρίλιο θα φέρει καινούρια πρόταση και σα ερωτώ μόνο του θα το εκπονήσει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα και μόνο του θα το εισαγάγει και θα το εφαρμόσει ή μήπω το έχει συζητήσει ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Μάρκχαρτ τα είπε αυτά. Ευχαριστώ. Φεστ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σότερ για την παρουσίασή σας. Έχω μια προσωπική ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά από την προφορά σας, εσείς είστε Άγγλος και μάλλον επίκειται το Brexit. Αυτό τι σχέση έχει με τη δική σας θέση και τους κανόνες για την επανεκατάσταση, τη μετεγκατάσταση και τη μετανάστευση. Αν η χώρα σας ε, πια μετά το Brexit δεν θα ενέχεται. Εσείς κάνετε εδώ πολιτική για το μέλλον, αλλά η ίδια σας η χώρα μάλλον θα εξαιρεθεί από αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αν ανησυχούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αφήξεις, μήπως να σταματήσουμε να διευκολύνουμε τους πολέμους και την αλλαγή καθεστώτων για να μην ε, φεύγουν οι πρόσφυγες. Η μόνη κρίση εδώ είναι η ανθρωπιστική κρίση των θυμάτων των πολέμων αυτών. Έχω δύο ανησυχίε. Σωστά είπατε ότι ανησυχείτε και εσεί βαθιά για την κατάσταση στη Λιβύη. Ηρωνικό ήταν αυτό που είπατε για την Μάλτα και ε, το θαύμα που έγινε στη μείωση εκεί των αφήξεων. Αλλά δεν είπατε τι συμφωνία έχει κάνει η Μάλτα με τη Λιβύη που ενδεχομένως να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όπου βασικά έχουν στη Λιβύη ο κόσμος σε ύδατα που ε, ήταν ε, λιβικά, ενώ η Λιβύη δεν είναι ασφαλές μέρος. Τι έγινε με την Κροατία. Ήταν την περασμένη ε, Πέμπτη, τελείως απαράδεκτη η ακρόαση που κάναμε για την κατάσταση στην Κροατία και ε, το πράσινο φως που θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κροατία για το Σέγγεν, ενώ ε, είναι ανδιαφυσβήτητη η παραβίαση του διεθνούς δικαίου με τις αποθήσεις που κάνουν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα και πώς αποφασίσατε να δώσετε ακόμα περισσότερα χρήματα στις κροατικές αρχές. Και τώρα έρχομαι στην ερώτησή μου, που είναι διπλή αναγνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν στοιχεία και αγωνίζεστε με ένα αξιοθρύνητο ε, οικονομικό μηχανισμό. Μάλλον μηχανισμό ελέγχου, συγγνώμη. Ε, οι Κροάτες ε, αρμοδίες αρχές λένε ότι όλα είναι εντάξει. Πού το ξέρετε, δεν έχουν πάει ούτε στα σύνορα. Τα χρήματα που στέλνετε εκεί μαζικά, πώς τα ελέγχετε τι κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς δαπανούν αυτά τα κονδύλια. Γιατί οι ΜΚΟ επιτόπου λένε ότι γίνουν στραβά αυτά τα πράγματα. Ε, το δικό μου συμπέρασμα είναι το εξή. Είτε ε, είστε τόσο ανίκανοι που δεν ξέρετε τι συμβαίνει, αλλά αυτό δεν το πιστεύω. Νομίζω μάλλον ότι όλα αυτά είναι μάλλον εσκεμένα. Ότι εσείς επιβραβεύετε χώρες που αποθούν κόσμο και ασφάλεια στα σύνορα, ακόμα και αν γνωρίζετε ποιο είναι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πώς παραβιάζεται. Θα ε, προσφύγετε επί παραβάση κατά της Κροατίας γιατί παραβιάζει το δικαίωμα ε, πρόσβαση στη διεθνή προστασία. Έχετε βάλει καθόλου όρους για τα ευρωπαϊκά χρήματα που στέλνετε εκεί και επιβραβεύετε ε, τις χώρες που αποθούν τον κόσμο. Η κυρία Μπούρκχαρτ. Αυτό ήταν το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σότερ. Έχω μια συγκεκριμένη διευκρινιστική ερώτηση. Μιλήσατε για την κατάσταση ε, τη μετρολογική, ότι έρχεται ε, χειμώνα. και στα kit, ε, στα hot spots και στους καταβλισμούς υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα για να προστατεύσει καλύτερα αυτά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης από το χειμώνα και να αποφευθεί ανθρωπιστική καταστροφή. Και δεύτερη ερώτηση. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα, διότι υπάρχουν επιτόπου κάποιοι δήμοι και κοινότητες που για διάφορους λόγους δεν ε, μπορούν να επομιστούν αυτό το βάρος. Και τι θα γίνει τώρα που έρχεται η χειμώνας, ο κόσμος είναι στα δάση, στα Βαλκάνια ε, και χάνει τη ζωή του θα περιμένουμε και άλλους θανάτους και αυτή την ανθρωπιστική κρίση που μπορούμε να την αποφύγουμε. Ευχαριστώ κύριο Σμέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά που παρουσιάσατε την πρόοδο που επετεύθη. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια με τις διαφωνίες στο Συμβούλιο μέσω, μέσω πρόθεσμα. Η συμφωνία με τη Μάλτα, η συμφωνία της Μάλτας μάλλον. Μόνο λίγες χώρες έχουν υπογράψει. Αφορά δεκάδες ανθρώπους που διασώζονται στη θάλασσα. Ερώτηση. Τι φιλοδοξίες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να προχωρήσουμε στο πλαίσιο της Μάλτας και για αποβιβάσεις και μετεγκαταστάσεις τι προβλέπετε και πώς θα συμμετάσχουν και άλλα κράτη-μέλη στο όλο σύστημα. Δεύτερη ερώτηση. Τα χρήματα. Τα χρήματα που στέλνουμε σε τρίτες χώρες στα πλαίσια συνεργασιών. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να παρακολουθήσετε συστηματικά πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται. Και για την πρόσφατη κατάσταση στην Τουρκία προβληματίζομαι. Η Τουρκία ήδη μετακινεί προς την ασφαλή ζώνη σύρους πρόσφυγες. Μήπως χρησιμοποιεί δικά μας χρήματα για να το κάνει αυτό, ελπίζω όχι. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι τα χρήματά μας δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για να επαναπροωθεί τους Σύρους πρόσφυγες ξανά πίσω στη Συρία. Ευχαριστώ κύριε Κούνσε. Κούνσε. Κούνκε. Κούνκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Σότερα. Η συνεργασία στο πλαίσιο του Σέγγεν στηρίζει συγκεκριμένες διαδικασίες και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά αυτοί οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα όντα στα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα μετανάστευσης. Ποια είναι η απόψή σας. Η κατάσταση σύνορα της Κροατίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τι γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Είναι τεκμηριωμένο αυτό. Αυτό είναι αποδεκτό. Ή μήπω είναι λόγος να παγώσει η συμμετοχή της Κροατίας στο σύστημα Σέγγεν. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση. Κύριε Διευθυντά, κύριε Σότερ, ευχαριστώ καταρχάς για τις εξηγήσεις σας και την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη βασίζεται και στην ερώτηση της κυρίας Αμπίρ Ελσαλάνη και της κυρίας Κούνε. Πόσοι άνθρωποι, ποιες είναι οι ροές ανθρώπων στη Βοσνία Ποια είναι οι συνθήκε ε, διαβίωσής τους στου καταβλισμούς εκεί. Δεύτερη ερώτηση. Δεν μπήκατε σε λεπτομέρειες σε κάτι άλλο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Συντονισμό μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου. Αν υπάρχει σταδιακή εναρμόνιση αυτών. Τι κάνετε ούτω ώστε σταδιακά να υπάρχουν κοινέ επαγγελματικέ πρακτικέ που ακολουθούνται και να υπάρχει συνοχή. Είναι και θέμα ανθρώπου να από ένα κάτω μέλο σε άλλο κάτω μέλο στα πλαίσια τη συνθήκη του Δουβλίνου. Λοιπόν, πάνω σε αυτό τι γίνεται. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Κίνγκ πρέπει ήδη να καταφθάνει. Μπορείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε, να περιοριστείτε σας παρακαλώ. Μπορείτε να συνοψίσετε. Να δώσετε απαντήσεις στις ερωτήσεις στο επόμενο δεκάλεπτο και θα ζητήσουμε από τον Επίτροπο Κίνγκ να περιμένει ένα δεκάλεπτο, αλλά όχι παραπάνω. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Λέει και ο Σότερ. Ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Και ευχαριστώ και για τι ερωτήσει σα. Ορισμένε δεν είναι και τόσο εύκολε. Ε, ακούω πολλέ ερωτήσει από διαφορά πρίσματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Πάντω θα προσπαθήσω ε, να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Έγιναν πολλές ερωτήσεις για το θέμα τη συνεργασίες με τρίτες χώρες ε, από διάφορες οπτικές γωνίες. Κάποιες ε, θεωρούν ότι είναι συμφωνίε, συμφωνίες, ε, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για συμπράξει. Πρέπει να είμαστε σαφεί Πρέπει να συζητούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Οποιαδήποτε λύση για να έχουμε να δώσουμε μια βιώσιμη συνολική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις που είναι περίπλοκες, που είναι δύσκολες, σημαίνει να φτάνουμε σε συμφωνίες, σε συμπράξεις με τρίτες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ε, απαρνηθούμε τις αξίες μας, τις αρχές μας, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορούμε όμως να φτάσουμε σε συμφωνίες με τρίτες χώρες και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους μπορούμε να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις για τις επιστροφές. Το χρειαζόμαστε αυτό για να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις επιστροφές που δεν είναι ικανοποιητική, διότι κάποιος ε, είπε πώς θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ οικονομικών μεταναστών και ανθρώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Αυτού που πρέπει να του προστατεύσουμε, να του προστατεύσουμε. Αυτοί όμω που είναι οικονομικοί μετανάστε και δεν θα πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να μπορούμε να βρούμε ε, έναν τρόπο στο μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να επιστρέψουν. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Δημιουργώντα αυτέ τι ε, συμπράξει λοιπόν, τι ε, εταιρικέ σχέσει, διακανονισμού για τι επιστροφέ, εθελοντικέ επιστροφέ επίση. Έχουν γίνει αρκετέ εθελοντικέ επιστροφέ και συνεργαζόμενοι με τους διεθνούς, διεθνείς εταίρους μας όπως ο IOM ε, έχουμε πακέτα επανένταξης έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες προέλευσής τους. Είναι δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Θα πρέπει να πλαισιώσουμε καλύτερα και την πολιτική ανάπτυξης ε, για να μας απασχολούν τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό αυτά, αυτό και για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την ευρύτερη συγκυρία. Ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε συμπράξεις μέσω ε, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, μέσω πιλωτικών προγραμμάτων. Τέθηκε ένα ερώτημα για τα πιλωτικά προγράμματα. Είναι σημαντικά αυτά τα προγράμματα, υπάρχουν, είναι μικρής κλίμακα αυτή τη στιγμή, αλλά η πρόθεσή μας ε, είναι, και υπάρχουν χρήματα γι' αυτό, να υπάρξει έτσι μία αναβάθμιση. Ε, Πολλά κρατημέλη συμμετέχουν, ε, η Ισπανία με το Μαρόκο, αλλά και άλλα παραδείγματα. Ε, είναι πιλωτικά προγράμματα βέβαια, είμαστε σε πρώιμο στάδιο ακόμα, αλλά μας δείχνουν ένα δρόμο. Και αυτό είναι και προς όφελος ε, της χώρας προέλευσης, διότι μεταδίδουμε και κάποια εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής που μπορεί να είναι χρήσιμη, πολύτιμη όταν οι ενδιαφερόμενοι επιστρέφουν. Ε, νομικές λοιπόν ε, νόμιμες οδοί, συνεργασία, ε, πιλωτικά προγράμματα. Μαζί βεβαίως με τις συμφωνίες επανεισδοχής ε, και τους, και του διακανονισμούς. Και αναφέρθηκα προηγουμένω στην βελτίωση τη κατάσταση με τι επιστροφές. Η δυνατότητα που θα, γίνεται, θα δίνεται στο μέλλον στα πλαίσια του νέου κώδικα θεωρήσεων που θα τεθεί σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2020 και θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε, υπάρχουν αυτά. Ε, κάποιοι αναφέρθηκαν τον όρο κρίση που χρησιμοποίησα. Ακούστε, εγώ αναφέρθηκα στην κρίση ε, ε αναφερόμενο στο παρελθόν, σε ό,τι φορά στον αριθμό αφήξεων. Ε, δεν λέω ότι οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή αιτιολογούν τον όρο κρίση. Οι αφήξει αυτή τη στιγμή βεβαίω δεν πρέπει να μα κάνουν να ευσυχάζουμε, διότι η κατάσταση είναι ασταθή. Είδαμε ότι αλλάζουν ε, οι ροέ από τη μία οδό προ την άλλη. Ε, έχουν πολλές δύσκολες καταστάσεις σε πολλές περιοχές στον κόσμο, στη Λιβύη, στη Συρία ε, και βλέπουμε πώς, ε, πώς ασταθής είναι η κατάσταση. Η πίεση υπάρχει, δεν υπάρχει λοιπόν ε, περιθώριο φυσικασμού. η αλήθεια είναι ότι η λέξη κρίση δεν αιτιολογείται με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ. πρέπει όμως να μάθουμε από το παρελθόν. Να μάθουμε από την πραγματική κρίση πριν από μερικά χρόνια και θα πρέπει γι' αυτό να θεσπίσουμε ένα καλύτερο σύστημα. Και μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί θεωρούν ότι η κατάσταση ε, βρίσκεται σε αδιέξοδο, είναι κολλημένη, εν πάση ε, στο μέλλον όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξεκινήσει, ε, να οικοδομήσει μια νέα προσπάθεια στα πλαίσια αυτού του πακέτου. Δεν έχουμε άλλη αλλακτική. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και αυτή είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέθηκε και ένα συγκεκριμένο ερώτημα ε, για, τις, ε, για την επανεγκατάσταση. Δόθηκαν κάποια αριθμοί μάλιστα. Η επανεγκατάσταση είναι πολύ σημαντική, αυτό το γνωρίζουμε. Ε, η, κράτη, τα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα έχει πετύχει μια σειρά από πράγματα και αυτό αποτελεί επίτευγμα, θετικό στοιχείο. Όπως άλλες, ενώ άλλες χώρες ε, ε, στον κόσμο επιστοδρομούν σε ζητήματα πανεδοχής, εμείς βελτιωνόμαστε. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτές τις νόμιμες οδούς, ε, παρά τις παράτυπες και όχι τις παράτυπες που ουσιαστικά τροφοδοτούν τα, τα δίκτυα λαθρεμπόρων αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα κατάσταση. 15 κρατημέλη έχουν πει ότι θα δώσουν, θα προσφέρουν πάνω από 50.000 θέσεις και ω 7 Οκτωβρίου 2019 39.000, 78% δηλαδή από αυτό το σύνολο, αυτέ τι 39.000 θέσει έχουν πληρωθεί, έχουν γίνει επανεγκαταστάσει λοιπόν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στι 50.000, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, δίνουμε κάποιου μήνε παραπάνω έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για αυτό το σκοπό. Πλησιάζουμε λοιπόν τι 50.000 ε, οπότε αυτό μα δημιουργεί μια κάποια ικανοποίηση σε ό,τι αφορά τι έχουμε κάνει με την επανεκατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα πιο σταθερό σύστημα. Ε, γι' αυτό είναι σημαντικό το πλαίσιο επανεκατάστασης να θεσπιστεί. Ε, είναι πολύ καλό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εργαστεί έτσι ώστε αυτή η πρόταση να φτάσει σχεδόν σε, σε ολοκλήρωση. Εμείς ελπίζουμε να εγκριθεί σύντομα. Ε, δεν μου αρέσει εδώ να μιλάω για όρους, αλλά πρέπει να, να σκεφτούμε στρατηγικά όταν μιλάμε για επανεγκατάσταση. Πάρτε το παράδειγμα του μηχανισμού transit. Θα πρέπει να δούμε πού θα επικεντρώσουμε την προσοχή των κρατών μελών όταν έχουμε ε, κενώσεις από τη Λιβύη προς τη Ρουάντα ή στον Νίγηρα πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον ε, μηχανισμό επανεγκατάστασης για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις στρατηγικές στρατηγικά συμφέροντα ε, στα σημεία δηλαδή που είναι προτεραιότητα, προτεραιότητα για μας και νομίζω ότι εδώ έχουμε μια χρήσιμη και βελτιωμένη ένα βελτιωμένο τρόπο για να το κάνουμε αυτό ένα άλλο ζήτημα που ανέρχεται συχνά είναι αυτή η ανησυχία για τις αποθήσεις, τα pushback ε, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κροατία. Ακούστε, δεν θέλω να επαναλάβω τη συζήτηση αυτή για την προσχώρηση στο Σέγγεν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσω για τα pushback και τις αποθήσεις οποιαδήποτε απόθεση, οποιαδήποτε αίτημα απόθεση, οποιαδήποτε μάλλον ε, ε καταγγελία απόθεση, είναι κάτι το παίρνουμε πολύ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχει μια αξιολόγηση προσω, ε, προσωπική τη κάθε της ασύλου. μιλάτε βεβαίως για την εφαρμογή του, του κεκτημένου ε, της Ένωσης. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά πρέπει να μπείτε και στη θέση μα. Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε εκεί τη στιγμή που λαμβάνει η χώρα η απόθεση και να γνωρίζουμε να έχουμε τα στοιχεία, τα αποδεικτικά ότι όντω έγινε, έγιναν. Εμείς εξετάζουμε, δίνουμε συνέχεια στις καταγγελίες που υπήρξαν σε ό,τι αφορά την Κροατία. Ένας άνθρωπος του DG Home πήγε στην Κροατία και ερεύνησε το ζήτημα, όμως σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, τα αποδεικτικά, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο να το συμπεριλάβουμε σε μια διαδικασία επί παραβάση. Πάντως, οποιαδήποτε καταγγελία την παίρνουμε πολύ σοβαρά και συνεργαζόμαστε με τα εν λόγω κρατημέλη, έτσι, έτσι λειτουργούμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, πρέπει να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές. Σας, σας διαβεβαιώ ότι δίνουμε συνέχεια στα θέματα αυτά, τα παρακολουθούμε. Η συμφωνία της Μάλτας τώρα και το θα γίνει από εκεί πέρα. Ε, ναι, πρέπει να κλείσω. Βέβαια μου τέθηκαν και ερωτήματα. Πώ θέλετε, Πρόεδρε. Κάντε ό,τι μπορείτε, λέει ο Πρόεδρο, διότι περιμένει ο Επίτροπο. πρέπει να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε το χρόνο. Ναι, θα απαντήσω για τη Μάλτα μόνο. Ε, ως Κομισιόν εμείς θα θέλαμε όσο γίνεται περισσότερα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων κρατών μελών στην οποία αναφέρθηκα. Αυτή η συμφωνία είναι εξαιρετικά θετική διότι αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετική προοπτική ε, τα έχουν βρει. Και αυτό ε, μας δίνει μια θετική ένδειξη για το πώς μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν σημαντικό και η Κομισιόν έκανε προσπάθεια το καλοκαίρι να διευκολύνει τις ε, αποβιβάσεις, αλλά πρέπει αυτές οι αποβιβάσεις ε, ε, είτε γίνεται στη Μάλτα, στην Ιταλία, ότι αυτές οι χώρες δεν θα μείνουν μόνες. Η Γερμανία, η Γαλλία ήταν εκεί, υπήρχαν και άλλα κράτη-μέλη όμως. Αυτό το οποίο είναι ελπιδοφόρο με τη δήλωση αυτή είναι η περαιτέρω σαφήνεια που υπάρχει σε ό,τι αφορά την προβλεψιμότητα. Και η Κομισιόν ε, το παρακολουθεί αυτό μετά την ε, έγκριση της δήλωσης αυτής. Ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη αλλά και με άλλους φορείς για να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη συνεργασία και με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, την Frontex, την EASO, για να μπορέσουμε με πρακτικό τρόπο να δείξουμε ότι η ελληνική λειτουργεί μπορεί να γίνει αυτό αποτελεσματικά και δίκαια μεταξύ κρατών μελών και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα πάνω στο οποίο θα βασιστούμε όταν θα γίνει αυτή η συζήτηση σύντομα, ελπίζω, για το, ευρωπαϊκό, για το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Αυτά και ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να είμαστε ευγενικοί και απέναντι στον επόμενο καλυσμένο τον κύριο Κίνγκ. Λοιπόν, όχι διαλύματα, παρακαλώ, και διακοπές και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση συνεχίζουμε ένα κτίριο λάκτισμα για το επόμενο θέμα. Δεν κάνετε φασαρία τώρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, Έχουμε και πάλι την τιμή να καλωσορίζουμε εδώ στο Προεδρείο ως προσκεκλημένο ομιλητή μας τον Επίτροπο κύριο Κίνγκ. Μια χαρά σας βλέπω. Βιαστήκαμε να σας αποχαιρετήσουμε κύριε Κίνγκ, κύριε Επίτροπε και έρχεστε ξανά και ξανά. Ε, να μας μιλήσετε για αυτό το σημαντικό θέμα της 20ης έκθεσης πρόοδου για την Ένωση Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πρόοδους στον τομέα αυτό και έχει θέσει και προτεραιότητες που απαιτούν κάποια δράση σύμφωνα με την τρέχουσα ακόμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να ακούσουμε από εσά λοιπόν κύριε Επίτροπε τα βασικά στοιχεία αυτής της 20 η έκθεσης για την Ένωση Ασφαλείας. Έκθεση προόδου επαναλαμβάνω. Γίνονται προσπάθειες για μια νέα στρατηγική ασφαλείας, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή μα έχει τονίσει ότι η νέα Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει ε, ε, την ε, εργασία της και τις αναφορές αυτές τις διαρθρωμένες. Επίσης γνωρίζουμε όμως ότι ο επόμενος επίτροπος δεν θα έχει, μάλλον δεν υπάρχει χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχωριστό και εντάσσονται στα θέματα εσωτερικών υποθέσεων. Δεν υπάρχει δικό επίτροπος ασφαλείας με αποκλειστική αρμοδιότητα και τέτοιο χαρτοφυλάκιο. Έχουμε λοιπόν το προνόμιο να ακούσουμε την παρουσίασή σας, κύριε Κίνγκ. Σας δίνω το λόγο. Σας παρακαλώ για τα επόμενα 15 λεπτά. Έχουμε προγραμματίσει χρόνο μέχρι τις 5.30. Θα έχουμε χρόνο και για συζήτηση και μην ανησυχείτε, ετοιμαστείτε. Το λόγο έχετε κύριε Κίνγκ εσείς. Ευχαριστώ Προέδρε, καλησπέρα. Αξιότιμα μέλη, συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαι εδώ για μία ακόμη φορά περαιτέρω δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα της ε, Ένωσης Ασφαλείας και τα θέματα ασφαλείας, όπως είπε και ο Πρόεδρο και παρατηρήσατε. Είχαμε σύμπτωση γεγονότων τέτοια που είμαι επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εδώ, λίγες εβδομάδες ακόμα. Θα με ανεχθείτε, αλλά είστε βέβαιοι, και το εννοώ αυτό. Είναι σαν εκείνες τις, τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 που λέγανε ότι φεύγουν και ξαναρχόταν. Το εννοώ όσο είμαι εδώ, μέχρι τελευταία μέρα θα εργάζομαι στο ρόλο μου από αυτού του θέματος. Τα θέματα αυτά είναι σημαντικά. Τι συζητάμε σήμερα, την 20η έκθεση για την ασφάλεια στην Ένωση. Την διάβασα όπως και άλλοι. Ε, είναι ογκώδης έκθεση, πολύ βαριά, αλλά είναι και σημαντική δυνατότητα να αναθεωρήσουμε αυτά που πετύχαμε πρόσφατα, τι πετύχαμε από κοινού αλλά να δούμε και ποιε προτεραιότητε πρέπει να έχουμε στο μέλλον, γιατί χρειάζεται και κατεπίγουσα δράση σε κάποιου τομεί. Τα τελευταία χρόνια μαζί είδαμε τη φύση των απειλών. Αλλάζει η φύση τους συνέχεια και αυξάνεται η δύναμή του, Ανταποκριθήκαμε προσπαθήτας να δημιουργήσουμε αποτελεσματική ένωση ασφαλεία. Σημειώσαμε πρόοδο θεωρώ, αλλά πολλά απομένουν να γίνουν και προσβλέπω στη σχετική συζήτησή μα. Τρομοκρατία. Όσον αφορά την τρομοκρατική απειλή, κλείσαμε τους χώρους για τους τρομοκράτες, να μην παρακινηθούν με ενός κανόνε, του δυσκολεύουμε την πρόσβαση, εκρηκτικά, πυροβόλα όπλα, χρηματοδότηση Φερρυπίν, όλα αυτά καλύπτονται, ανταλλαγή πληροφοριών αυξήθηκε, με μέτρα προς βελτίωση διελειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μας, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση υφισταμένων πληροφοριών και να καλύψουμε τυχόν κενά και τυφλά σημεία που υπήρχαν. Προσπάσαμε να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, υποστηρίξαμε εκείνου που εργάζονται επί τόπου, στι κοινότητε με γι' αυτό, ανταλλαγή των πρακτικών. Δημιουργήθηκε συνεργασία με τι πλατφόρμε του διαδικτύου και προτείναμε νέου κανόνε για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματο του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυξήσαμε την αντοχή μα κατά των επιθέσεων με σχέδια δράση να υποστηρίξουν προστασία δημοσίων χώρων και να βελτιώσουμε τη δυνατότητά μα να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάποια μέσα που χρησιμοποιούνται βιολογικά, χημικά, ραδιολογικά, διάφορους, διάφοροι φορείς, η Europol και η Eurojust, υποστήριξαν τα κράτη-μέλη για να πολεμήσουν καλύτερα την τρομοκρατία, το έγκλημα, το κυβερνοέγκλημα Πρόσφατο παράδειγμα που έδωσε και την άλλη μέρα, την άνοιξη φέτος η Europol και η Eurojust υποστήριξαν τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Ηνωμένε Πολιτείε για να μειώσουν, να συντρίψουν την αγορά του Dark Net, τη Wall Street Market, τη δεύτερη αγορά, όπου εκεί μπορούσαν να εμπορεύονται κλεμμένα στοιχεία, ψευδή έγγραφα, διάφορα επιβλαβή προγράμματα, ε, ναρκωτικά. Δείχνει αυτό τι προβλήματα έχουμε ε, στον κυβερνοχώρο νέα μέσα αναπτύσσονται, πρέπει και εμεί στην ανταπόκρισή μα να αναπτυχθούμε. Έχουμε νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια, αυξήσαμε την τυχή μα, είναι πιο δύσκολο να μα επιτεθούν τώρα και αν συμβεί το χειρότερο, να μπορούμε να ανακάμψουμε το ταχύτερο δυνατό. Ενισχύουμε τα μέτρα αποτροπή μα στο διαδίκτυο, αυξάνονται οι πιθανότητε να συλληφθούν οι επιτιθέμενοι και να τιμωρηθούν και υποστηρίζουμε και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τη δική του άμυνα. Έχουμε εργαλειοθήκη για την κυβερνο και θέλουμε να έχουμε και πλαίσιο ε, πιστοποίησης για να αυξήσουμε τα πρότυπα κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχαμε αύξηση στα προβλήματα τα σχετικά με απειλές που κινούνται μέσω του κυβερνοχώρου, κυρίως παραπληροφόρηση στον πολιτικό χώρο που έχει σαν στόχο τις δημοκρατικές μας διαδικασίες και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Συζητήσαμε λοιπόν το θέμα και δημιουργήσαμε αντίμετρα πάνω σε αυτό, σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση για να εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε συντονισμένε εκστατείε παραπληροφόρηση. Κινητοποίησαμε την κοινότητα εκείνων που ελέγχουν την πραγματικότητα, τα στοιχεία, ερευνητέ κινούνται σε αυτό. Συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τι εκστατείε παραπληροφόρηση. Πιέσαμε επίση τι μεγαλύτερε πλατφόρμε του διαδικτύου να ενταχθούν σε έναν κώδικα δοντολογικό εστιαζόμενοι επί των προβλημάτων της πολιτικής παραπληροφόρησης και λογοδοτούν αυτοί αν θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Εδώ και τη βδομάδα δημοσίευσαμε την πρώτη έκθεση αυτοαξιολόγησης εκείνων που είχαν υπογράψει το δοντολογικό κώδικα των διαφόρων πλατφορμών που καθορίζουν πολιτικές διαδικασίες και δράσεις που δρομολόγησαν για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους ευπρόσδεκτη η δέσμευση των ε, διαδικτυακών πλατφορμών να επεξεργαστούν το θέμα, να γίνουν διαφανέστερες, αλλά ειλικρινά ποικίλει η πρόοδος μεταξύ των συμβαλωμένων μερών, μεταξύ στοιχείων και χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να εξετάσουμε ποιο αντίκτυπο πραγματικό έχουν τα αυτορυθμιστικά μέτρα τα οποία εφάρμοσαν τον τελευταίο χρόνο και πρέπει να επανεξετάσουμε τους μηχανισμούς για ανεξάρτητο έλεγχο. Το ότι αυτόματη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση υπάρχει και είναι αυτομάτου χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι σε όλου του τομεί θα πρέπει να εργαστούμε όσον αφορά τον κώδικα. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτό ότι θα ισχύει για πάντα. Λοιπόν, τελικό βήμα αυτή τη ετήσια ε, διαδικασία είναι η επίσημη αξιολόγηση που θα γίνει τέλο Ιανουαρίου μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις με ανεξάρτητους εμπειρογνωμόνες και με τα κράτη-μέλη της της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αρχές επομένου έτους. Αν τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δείξουν ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, τα συζητήσετε αυτά, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εξετάσουμε τι δεν γενέστε ίσως περαιτέρω δράσεις και ενδεχομένω κάποιο κανονισμό. Ταυτοχρόνως θέλαμε να εξασφαλίσουμε τις ψηφιακές κρίσιμες υποδομές σε σχέση με τα μελλοντικά δίκτυα 5G, πέμπτης γενιάς, 5G. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να προστατευτεί, γιατί θα είναι σημαντικό για επικοινωνία, για οικονομία και για την κοινωνία το 5G. Άρα πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό. Δεν είναι μόνο η, η ποιότητα των διασυνδέσεων, αλλά επίσης και εκείνος που παρέχει υπηρεσίε. Δηλαδή, ο εξοπλισμός 5G πρέπει να αξιολογείται διεξοδικότατα, πιο διεξοδικά από ό,τι πριν, όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για το δίκτυο 5G και οι πρακτικέ για την κυβερνοασφάλεια και πιθανότητα ο προμηθευτή να υπόκειται σε παρέμβαση από τρίτη χώρα. Δεν χρειάζεται να το πω λεπτομερώ. Εδώ και μερικέ εβδομάδε, 28 κράτη-μέλη με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Κυβερνοασφάλεια δημοσίευσαν μια έκθεση σχετικά με τη συντονισμένη εξολόγηση κινδύνου Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την κυβερνοασφάλεια δωμέα στον τομέα 5G και το επόμενο βήμα θα είναι μέχρι τέλο του έτου ξανά μαζί με τα κράτη-μέλη να εκπονηθεί σειρά μέτρων προσλήψη εθνικό ή συλλογικό για τη διαχείριση και μείωση των κινδύνων. Σε όλα αυτά Θέλουμε να αξιολογήσουμε, να ακολουθήσουμε προσέγγιση βάση κινδύνων. Δεν έχουμε στόχο συγκεκριμένη περιοχή, συγκεκριμένο προμηθευτή, αλλά τούτου λεχθέντο υπογραμμίζαμε πάντα ότι με αυτή την επιφύλαξη για την μείωση αρνητικών αποτελεσμάτων κάποια προϊόντα και υπηρεσίε οι προμηθευτέ ίσω να δημιουργήσουν προβλήματα που ίσω θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό λοιπόν στους διάφορους τομείς καταφέραμε να προχωρήσουμε και σημαντικά μάλιστα την τελευταία τριετία αλλά υπάρχουν πολλά που να γίνουν αυτές οι απειλές δεν απομακρύνονται το συγκυβερνοχώρο, την παραπληροφόρηση, την τρομοκρατία ε, κυρίως πέρα από την απειλή που δημιουργείται από τους τζιχαντιστές και τη τζιχαντιστική τρομοκρατία βλέπουμε μια αύξηση σε, βία από, την, από τον ακροδεξιό εξτρεμισμό και ε, επιθέσεις όπως αυτή, αυτή που σημειώθηκε στο Χάλε πρόσφατα. Θα πρέπει κατεπηγόντως να πετύχουμε μια συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Οι προτάσεις δεν καλύπτουν μόνο τζιχαντιστικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες εξτρεμιστικές εκφράσεις που αναλογούν σε τρομοκρατικές πράξεις. Θέλουμε να δώσουμε ασφάλεια δικαίου και θέλουμε ασφαλή μέτρα για να αποφύγουμε τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, εξασφαλίζοντα ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση με την ελευθερία του λόγου και τη ενημέρωση. Χαίρομαι που γίνεται συζήτηση στα πλαίσια τριμερού διαλόγου με εσά και με το Συμβούλιο. Έγιναν αυτές οι συνομιλίες αρχές Οκτωβρίου. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάκη και όλους του κοιόδη συζητητέ για τι προσπάθειε που κατέβαλαν και ελπίζω ότι μαζί θα μπορέσουμε γρήγορα να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο. Υπάρχουν και άλλα εκρεμή θέματα, νομοθετικέ προτάσει που χρειάζονται γρήγορη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Χαίρομαι που υπάρχει σχέδιο εκθέσεω για τι ηλεκτρονικέ αποδείξει. Δεύτερον, για, ευρωπαϊκή, ε, για ένα κέντρο δίκτυο, η ευρωπαϊκή τεχνολογία και κέντρα συντονισμού για την χρήση ασφαλείας ε, στον ε, κυβερνοασφάλεια σε όλους τους τομείς βιομηχανικής παραγωγής. Μετά θέλουμε συστήματα ισχυρά και ευφυή για τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, κυρίως οι τεχνικές αλλαγές της νομοθεσίας για το αιτίας. Αυτές οι προτάσεις ε, είναι σημαντικές όλες αυτές για να έχουμε μια ένωση ασφαλείας. Εν γέννη λοιπόν, και εστιάζομαι για λίγο πάνω σε αυτό, η απειλή που προέρχεται από τζιχαντιστική τρομοκρατία δεν έχει φύγει με το θάνατο του Αλμπαγκδάντι, δεν θα πρέπει να αισθανθούμε χαλαροί πέρα από, την, από το πρόβλημα αυτοριζοσωτικοποιημένων ε, ανθρώπων πριν να δούμε τι γίνεται στις φυλακές κάποιοι που έχουν περάσει κάποια ποινή στη φυλακή λόγω τρομοκρατίας ή έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί στη φυλακή τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε πρόβλημα με τους ξένους μαχητές τα γεγονότα στη Συρία δεν διευκολύνουν την κατάσταση Λοιπόν, φυλακισμένα μέλη του Ντάις που το έσκασαν, αυτή η διαφυγή ίσως να έχει συνέπειες ασφαλείας σημαντικές για μας. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πλήρως την εφιστόμενο σύστημα πληροφοριών για να εντοπίσουν ξένους μαχητές όταν αυτοί διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα. Επίσης συνεχίζεται δουλειά όσον αφορά την χρήση πληροφοριών από τα πεδία της μάχης για να εντοπίσουμε και να διώξουμε ξένους μαχητές. Τούτου λεχθέντος πιστεύω ότι είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι σήμερα από ότι ήμασταν εδώ και κάποια χρόνια για να αντιμετωπίσουμε και να εντοπίσουμε μάλλον και να αντιταχθούμε σε εκείνους που ίσως αποπειραθούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη με πρόθεση ε, περαιτέρω βιοπραγιών κατά των συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζουν πλήρως μέτρα τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί όπως η πρόσφατη νομοθεσία περί διαλειτουργικότητα και η νομοθεσία για πρόδρομες ουσίες, για εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα. Εξακολουθούμε να επιδιώκουμε ε, αποτελεσματική εφαρμογή των συμπεριφανθέντων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο για εφαρμογή όπως το PNR, οδηγία για την καταπολέμηση των τρομοκρατών και την οδηγία, την προστασία ε, των δεδομένων, αλλά απομένουν κι άλλα να γίνουν για τις οδηγίες που αφορούν κυβέρνο έγκλημα, όπου αναφέρονται λεπτομερώς αυτές οι οδηγίες στην έκθεση. Επίσης, για την αύξηση της ασφαλείας μας, κάνουμε δουλειά. Δεν περιορίζεται αυτή μόνο στην Ευρώπη, συνεργαζόμαστε και με χώρες εταίρους ενεργά υποστηρίζουμε διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες στις προσπάθειες που καταβάλουν και αυτή Ένα παράδειγμα, να προσέξουμε, συμβάλλουμε οικονομικώς στο πρόγραμμα καταπολέμησης ταξιδίων του, ταξι, του να δίνει αντιτρομοκράτες να ταξιδεύουν. Ε, είναι κάτι που ενδιαφέρει πολλές περιοχές του κόσμου. Να εφαρμόζουμε την 2396 από το Συμβουλίου Ασφαλείας του 2017 που θα πρέπει τα κάτι με σύμφωνα με αυτά να απτύξουν τη δυνατότητα να επεξαργάζονται τα PNR. Όπως ξέρετε η πρωτοβουλία του ΟΗΕ καλύπτει τη Δυτική Αφρική. Η εφαρμογή ξεκίνησε στο Τόγκο, Γκάνα, Σιέρα Λεόνε ακολουθούν και πολλές άλλες χώρες. Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμβια, Μαυριτανία, Νιγηρία και Νίγηρας που ενδιαφέρονται διακαώζει το θέμα. Λοιπόν, το πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ταξιδιού των τρομοκρατών συνεπάγεται και άλλε περιοχέ όπου που ταξιδεύουν πολύ επιβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια, Νότια, Αφρική, κέρα Αφρική, Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία, ε, περιοχή Ειρηνικού ε, κλπ. Οπότε θα υποστηρίξουμε τον ΟΗΕ σε όλε τι προσπάθειε που καταβάλει. Τέλο, για τη Νέα Ζηλανδία. Μαζί με την έκθεση για την ασφάλεια στην Ένωση που διαβάζουμε σήμερα, έχουμε κάνει συστάσει στο Συμβούλιο για διοδότηση εντολή να ξεκινήσει πραγματεύσει με τη Νέα Ζηλανδία για ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων για καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματο και τη τρομοκρατία. Αυτό ακολουθεί το μοντέλο και έχουμε τα ίδια μέτρα διαφύλαξη για τα δικαιώματα όπω με χώρε προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή τη Βορειοαφρική, μέτρα που υθετήθηκαν το Δεκέμβριο του 2017. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη γι' αυτό. Είναι μια μηδέα ευκαιρία και για τι δύο χώρε να αυξήσουμε συνεργασία όσον αφορά τα θέματα ασφαλεία με τη Νέα Ζηλανδία. Επεσκέφθη η Νέα Ζηλανδία το μήνα Ιούνιο. Ξανά κατέστη σαφέ ότι η Νέα Ζηλανδία έχει την ίδια άποψη όπω και εμεί. Αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια και στενότερη συνεργασία θα ήταν επικοδομητική και για μας αλλά και για αυτούς. Ήδη συνεργαζόμαστε με τη Νέα Ζηλανδία όσον αφορά τη, το, τη χρήση του διαδικτύου για απειλέ, παραπληροφόρηση και 5G. Μελλοντική συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία για προσωπικά στοιχεία την καταπολέμηση τρομοκρατίας θα επεκτείνει συνεργασία σε σημαντικούς τομείς όπως καταπολέμηση κυβερνοεγκλήματος, εκμετάλλευση των παιδιών, εξαλικής εκμετάλλευση των παιδιών και τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και δυστυχώς αυτό το ξαναείδαμε μετά την επίθεση στο Christchurch ε, τον Μάρτιο φέτος. Τι δείχνει αυτή η συμφωνία, δείχνει ότι οι πιο στενοί μας σύμμαχοι, οι εταίροι μας που έχουν παρόμοια νοοτροπία μπορεί να είναι πολύ μακριά από εμά. γιατί εδώ μιλάμε για αξίες, δεν μιλάμε για γεωγραφική θέση και νομίζω ότι η σχέση μας με τη Νέα Ζηλανδία είναι ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα αυτού που λέω. Κλείνοντας λοιπόν θέλω να πω ότι είναι η πιο πρόσφατη έκθεση τη Ένωση Ασφάλεια, αλλά όχι τελευταία, όπω είπε και ο πρόεδρο εν είδη εισαγωγή, οι συνάδελφοι τη επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαν ότι θα βρουν έναν τρόπο συνέχιση του έργου αυτού και να συνεχίζουν να σα ενημερώνουν για τα θέματα αυτά, σχετικά με αυτά που κάνουμε στο τομείς αυτής, ίσως να μην υπάρχει ένα που θα είναι υπεύθυνο για την Ένωση Ασφαλεία με αυτό το χαρτοφυλάκιο στα χέρια του. Από ό,τι βλέπω ε, τις αποστολές που ανετέθησαν υπάρχουν διάφοροι που ασχολούνται με τα θέματα ασφαλεία για την Ένωση. Θα συνεργαστούν αυτοί αποτελεσματικά σε όλε τι προσπάθειε που καταβάλλονται μέσω συνεργασία, σε όλα τα επίπεδα επιτυχάνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και ανταποκρινόμαστε στι επιθέσει και τι απειλέ. Αυτό δεν θα αλλάξει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Now, let's open discussion. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Κίνγκ για να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτα οι συντονιστέ και μετά οι υπόλοιποι διακόπτη ο Πρόεδρος. Λοιπόν, να ακούσουμε το σύνολο των ερωτήσεων πρώτα και στο τέλος εσείς θα απαντήσετε. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Ματσόλα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε ακόμα εδώ μαζί μας. Αναμένουμε βεβαίως τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας, ιδιαίτερα στα ζητήματα δρομοκρατικής απειλής. Σας ευχαριστώ και για τη εισφορά σας σε μια καλύτερη, για μια καλύτερη αλλαγή πληροφοριών, έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τους τρομοκράτες και να προστατεύουμε τους συμπολίτε μας. Γνωρίζουμε ότι έχουν λάβει χώρα πολλές επιθέσεις οι επιθέσεις αυτές που μπορούσαμε να σταματήσουμε, να αποτρέψουμε, ε, δεν βρίσκονται ε, στην επικαιρότητα, δεν φτάνουν στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι όμως μια απειλή πολύ πραγματική, όπως είπατε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ανοιχτοί στο διάλογο και να ολοκληρωθεί και η νομοθεσία για το τρομοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές επιγραμμικά ε, μετά την επιστροφή επίσης των ξένων μαχητών στις οικογένειές τους όλα αυτά αποτελούν ενδεχόμενες απειλές. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και τις πληροφορίες που έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη και τρίτες χώρες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, την προπαγάνδα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο διαδίκτυο, γιατί συχνά αντιδρούμε πολύ αργά, παρόλο υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια από στο παρελθόν. Θα πρέπει να δώσουμε σφαιρικές απαντήσεις σε αυτά τα παγκόσμια προβλήματα. Ε, οπότε πείτε μας πώς μπορούμε να αναλύσουμε τη συνεργασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο Γνωρίζουμε ότι κάποια κράτη-μέλη ε, αντιδρούν, αντιστέκονται στι απόπειρε που γίνονται. Πώ μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη θα είναι πιο ασφαλή, τι μπορούμε να κάνουμε, ε, ποια στοιχεία τη εργαλειοθήκη μα ε, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να μην είμαι εδώ για τις απαντήσεις, αλλά θα το ακούσω από το web streaming. Δύο λεπτά περίπου, παρακαλώ, οι παρεμβάσεις, διότι ήδη το πρώτο σημείο μας καθυστέρησε και μετά έχουμε και την κοινή συζήτηση με συζητήματα που θα κάνουμε με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, οπότε παρακαλώ να μην ε, χαθεί χρόνος. Πάντως μου άρεσε που άκουσα μαλτέζικα από κύριο Κίνγκ. Ναι, ναι, βεβαίως, λέει ο πρόεδρος, πάντα προσπαθούμε ε, να σεβαστούμε ε, τα επιχειρήματα και το σκεπτικό ε, όλων των ομιλητών, αλλά παρακαλώ σε δύο λεπτά μέσα θα ήταν καλύτερο. Κύρια Ζίπελ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω γερμανικά εγώ για αλλαγή. Θυμάμαι ότι μετά τις εκλογές συναντηθήκαμε με τον Επίτροπο Κίνγκ που θεωρούσαμε ότι ήταν η τελευταία ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Για να δούμε μήπως ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις ε, ανάλογα με τις εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, κύριε Κίνγκ, κύριε Επίτροπε, στην αρχή ε, η παρουσίασή σας είπατε ότι το πρόβλημα αυξάνεται όλο και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα και την δρομοκρατία, αλλά κυρίως με την αύξηση της ακροδεξιάς βίας. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ακροδεξία είναι μεγαλύτερο πρόβλημα στο μεταξύ ε, σε πολλούς τομείς από τις άλλες μορφές της τρομοκρατίας. Τα κράτη-μέλη μας όμως ε, δεν ε, εστιάζουν τόσο πολύ την προσοχή τους σε αυτή τη νέα εξέλιξη και θα ήθελα να ακούσω παρακαλώ τη δική σας εκτίμηση. Επίσης τονίσατε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με την ψηφιοποίηση προφανώς, με τις ηλεκτρονικές επιθέσεις ή την παραπληροφόρηση ε, στο διαδίκτυο και αναφέρατε τη συνεργασία αλλά και την πίεση ε, προς τους παρόχους ε, να συνεργαστούν. Έχω λοιπόν την εξής ερώτηση. Στις κρατικές αρχές πόσο μεγάλη είναι η πίεση να δρούν αποτελεσματικά, γιατί καλή είναι η σερβερ να συνεργαζόμαστε, αλλά ε, εάν δεν έχουν οι, κρατικέ οι κρατικές αρχές τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνογνωσία, το προσωπικό, τότε ε, μπορεί ε, να υπάρξει ιδιωτικοποίηση ε, καθόλου χρήσιμη αυτής της υπηρεσίας. Και εδώ τα κράτη-μέλη έχουν κάποια κενά να καλύψουν. Ε, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο που έμεσα συνδέεται με το δικό σας τομέα αρμοδιοτήτων. Όταν μιλούμε για την εσωτερική ασφάλεια, έρχεται η απάντηση από τα κράτη-μέλη αντανακλαστικά ότι αυτό είναι θέμα του κάθε κράτης μέλους. Εάν έχω παρακολουθήσει όμως τις εκθέσεις προόδου σας, ε, είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα τα θέματα της εθνικής ασφάλειας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Πολλές φορές και η εθνική ασφάλεια είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, γιατί πολλά προβλήματα είναι διασυνοριακά. Ε, σε σχέση με αυτά λοιπόν έχει σημασία και τα νομικά μας συστήματα σταδιακά να ε, συμπλησιάζουν. Αυτό το βλέπω συχνά όμως όχι μόνο στους νόμους ασφαλείας και άλλο ότι έχουμε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα για να εφαρμοστούν. Τα ίδια ισχύει για τον οδικό χάρτη, για τα δικονομικά δικαιώματα. Ε, σας ερωτώ εσείς πώς το βλέπετε αυτό από τη σκοπιά της πολιτικής ασφαλείας. Όταν δεν εφαρμόζονται τα δικαιώματα αυτά, τα ε, δικονομικά, ε, αυτό μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και να μειώσει και τη δυνατότητα δράσης. Ε, και τις τελευταίες μέρες με θορύβησε πάρα πολύ αυτό που έμαθα, γιατί αυξάνεται η εισαγωγή ναρκωτικών, ιδιαίτερα κοκαίνης, που έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Και είναι πολλές οι οδοί μέσω των οποίων φτάνουν αυτά τα ναρκωτικά. Μπορεί η Frontex εδώ πέρα να κάνει ε, αποτελεσματικούς ελέγχους ή ασχολούνται με άλλα θέματα αυτό το καιρό οι αρμόδιοι οργανισμοί. Uh, Ευχαριστώ πρώτα να ευχαριστήσω και τον επίτροπο που είναι εδώ. Ε, ε, η σύγκριση η, σύγκριση, με τον Κρόιφ είναι προφανής γιατί και αυτός ε, συνέχεια έφευγε και όλο δεν έφευγε και έπαιζε το τελευταίο του μάτι πολλέ φορέ και ήταν και δημοφιλή στο τέλο. Όπω εσεί. Λοιπόν, ε, δυο τρει πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτέ οι ανταλλαγέ πληροφοριών ορισμένε φορέ ε, ε, είναι μια διαδικασία ρουτίνα όπου επαναλαμβάνουμε τα ίδια, ε, θέλουμε τα ίδια ερωτήματα και δεν φαίνεται να σημειώνεται κάποια πρόοδο ε, ουσιαστικ, σε ουσιαστικά ζητήματα. Ε, Βεβαίως έχουν γίνει πολλά πράγματα για την ενίσχυση της ασφάλειας ε, ε, από πλευράς καταστολής, αν θέλετε. Όμως ε, πρέπει επίσης να γίνει μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά την νομική προστασία των πολιτών, της δικλείδας ασφαλείας. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά έχουμε αποτύχει και το έχω πει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και ακούμε τα ίδια από την Κομισιόν κάθε φορά, αλλά βελτίωση δεν βλέπουμε. Ε, υπάρχει μια τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο όλος ιδιαιτέρως να νομοθετούμε ε, νομοθετήματα τα οποία δεν είναι ε, νομικώς διασφαλισμένα κείμενα, δεν θα έχουν πραγματική επιρροή. Το PNR, παραδείγματος χάρη, είναι το αγαπημένο μου θέμα εδώ και 16 χρόνια είχαμε την γνώμη του δικαστηρίου για τη συμφωνία με τον Καναδά και βεβαίω γνωρίζουμε ότι αυτό ισχύει και με, για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται απολύτω τίποτα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιπραγματευτούμε τη συμφωνία με του Αμερικανού. Το μόνο που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι αξιολογούμε την εφαρμογή τη υπάρχουσας συμφωνία. Η υπάρχουσα συμφωνία αποτελεί παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τόσο απλό είναι. Είναι παράνομος, παράνομη αυτή η νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να την αποσύρει. Αν ένας, όταν ένα πολίτη παραβιάζει τον νόμο, τιμωρείται. Και εδώ έχουμε να κάνουμε παραβίαση τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πού είναι οι κυρώσει, λοιπόν. Η Κομισιόν συνεχίζει ε, λες και δεν συμβαίνει τίποτα και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης θέσαμε ερωτήματα για τη συμφωνία με την Αυστραλία, ε, τον Καναδά. Ε, ζητήσαμε αποδεικτικά στοιχεία ε, για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του PNR και η απάντηση που λαμβάνουμε κάποιος προεδρεύει εδώ από πίσω θα τελειώσω βεβαίως ε, Όταν κάποιος μιλάει, λέει ο πρόεδρος, οι υπόλοιποι πρέπει να το σέβονται αυτό. Είναι τόσο απλό. Και έχει το λόγο αυτή τη στιγμή η κυρία Ιντεβέλτ. Ναι, θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Το μόνο που κάνει η Κομισιόν είναι να μας παρουσιάζει παραδείγματα για την επιχειρηματική ε, τη. Του χρόνου πρέπει να παρουσιάσετε την έκθεση αξιολόγηση για την οδηγία PNR. Πώ θα αποδείξετε, όχι απλώ να το λέτε, πρέπει να αποδείξετε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα αυτή τη μαζική αποθήκευση και χρήση δεδομένων PNR. Δεν έχω δει καμία απόδειξη εδώ και 16 χρόνια. Θα γίνει κάτι τελικά. Η κυρία Στρίκ έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Κίνγκ για την παρουσίασή του. Ποτέ μιλές ποτέ. Σας έχουμε ήδη ευχαριστήσει για αυτά που έχετε κάνει και σας ευχαριστούμε εκ νέου. Τώρα, η απόψη σας για την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας ε, και εγκληματικότητας, προφανώς και εμείς το τονίζουμε αυτό, δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί σε ό,τι αφορά την επιρροή από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό ε, στον δημόσιο χώρο μας, αλλά ε, ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε ότι τα μέτρα μας ε, πρέπει να συμμορφώνονται με το δικό μας κράτος δικαίου και τους κανόνες του. Ε, εσείς δώσατε έμφαση στην ανάγκη προστασίας του δημόσιου χώρου μέσω, πραγματικ... μέσω πραγματικής εφαρμογής ε, των μέτρων που έχουμε πάρει και μέσω μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει όμω να προστατεύσουμε και την ελευθερία έκφραση. Και αναρωτιέμαι ε, πώ βλέπει ο κύριο Κίνγκ την υποστήριξη των μέτρων ε, για τους δημοσιογράφους που διεξάγουν έρευνες. Ε, είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ε, θα τους προστατεύσουμε, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους, διότι σε αυτή την εποχή παραπληροφόρησης τους χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Για την κυβερνοάμυνα τώρα, βεβαίως ε, έχουμε τις εθνικές στρατηγικές, όμως ε, πρέπει αυτές οι στρατηγικές να σέβονται την ιδιωτική ζωή. Και συμφωνώ με αυτό που κυρία Ιντεβελντ, υπάρχει αυτή η νομολογία, ξανά και ξανά το δικαστήριο ήταν σαφές για τα όρια της παρακράτησης δεδομένων, Αναρωτιέμαι λοιπόν τελικά τι κάνει η Κομισιόν για να εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες, αλλά και οι εθνικές νομοθεσίες συμμορφώνονται με την ομολογία αυτή σχετικά με την παρακράτηση δεδομένων. Διότι αυτή πρέπει να είναι η βάση. Ακόμα συζητάμε βεβαίως ε, ποια είναι η ερμηνεία, αλλά νομίζω πως είναι πλέον σαφή τα πράγματα. Ποια είναι τα όρια δηλαδή ε, σε αυτήν την μαζική ε, διατήρηση δεδομένων. Τι κάνει επίσης η Κομισιόν να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των προσώπων, των ε, πολιτών που ενδεχομένως έχουν πληγεί από την τρομοκρατία ή και από μέτρα κατά της τρομοκρατίας και τέλος για τους μαχητές, τους τζιχαντιστές. Είναι αλήθεια ότι με τα τελευταία γεγονότα δεν έχει πάψει να υπάρχει απειλή γίνεται μια συζήτηση για τους ξένους μαχητές και τον επαναπατρισμό τους. Ε, γνωρίζω ότι η Κομισιόν λέει ότι είναι ένα εθνικό θέμα, είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν θα μπορούσε να έχει ένα συντονιστικό ρόλο ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε ό,τι αφορά τις, την, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ε, και να ασκήσουν διώξει στους πολίτες τους που έχουν ε, κάνει τρομοκρατικά εγκλήματα. Τι λέτε γι' αυτό. Ο κύριος Φέστ, έχετε εσείς το, το λόγο. Η κυρία Ινετφέλ δεν σέβεται όταν καταχράτε του χρόνου τους, τους υπόλοιπους βουλευτές. Και το ίδιο ισχύει και για τη δική σας ασέβεια, κύριε Λόπες Αγγιλάρ, που ανέχεστε αυτή την ασέβεια. Εν πάση περιπτώσει, η ασφάλεια ήταν προτεραιότητα ε, στη θητεία του Jean-Claude Juncker, αυτό το λέει και η αντίστοιχη έκθεση σήμερα. Αν δούμε όμως τα νέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2019, p News, εκεί λέει ότι το 2014 είχαμε ε, δύο ε, επιθέσεις με τέσσερις νεκρούς, τώρα είναι 24 αυτές με 13 νερούς ε, και, και άλλες 150 νεκροί και άλλοι για λόγους θρησκευτικού. Και ξέρουμε ότι 10 με 15 χιλιάδες παράνομοι μετανάστες φτάνουν στη Γερμανία, χωρίς χαρτιά, χωρίς ταυτότητες, χωρίς τίποτα. Και αν δεν το αλλάξετε, οποιαδήποτε καταπολέμηση τρομοκρατίας είναι χήμερα. Ε, και ε, οι τρομοκράτες που σκότωσαν τόσο κόσμο στον Πατακλά ε, ήρθαν από τη Γερμανία. Αυτό είναι πασιφανές. Γιατί δεν κάνετε τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ε, της πολιτικής του ξέφραγου αμπελιού των συνόρων που πρεσβεύει η κυρία Μέρκελ. Αυτή είναι η πύλη εισόδου της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και αυτή θα πρέπει να κλείσει επιτέλους. Δεύτερον, στην έκθεση ασφαλείας σας λέγεται ότι είναι προτεραιότητα η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτή δεν είναι ουρανοκατέβατη χρειάζεται αυτό οι μάμιδες, τζαμιά, διαδίκτυο, φυλάδια και βιβλία. Και όλοι γνωρίζουμε ότι κυρίως χρειάζεται χρήματα η ριζοσπαστικοποίηση και ξέρουμε και πριν είναι οι χρηματοδότες. Το κανάλι Άρτε, το γαλλογερμανικό, είχε κάνει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο βασικός χρηματοδότης είναι το Κατάρ αφενός και αφετέρου η Σαουδική Αραβία. Ούτε κουβέντα στην έκθεσή σας σχετικά απλώς γενικόλογα, σαφή ε, συνοθηλεύματα ε, και διατυπώσεις για παραπληροφόρηση και τα λοιπά. Δεν βοηθάει αυτό να καταπολεμήσουμε σε καμία περίπτωση τη ριζοσπαστικοποίηση. Και ρωτώ, αυτούς τους μουσουλμάνους χρηματοδότες της ε, ριζοσπαστικοποίησης, πότε θα τους αντιμετωπίσετε, πότε θα ακολουθήσετε το χρήμα για να λάβετε επιτέλους μέτρα να σταματήσετε αυτή τη χρηματοδότηση προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Φέστ, κοιτάξτε, το σχόλιο μου είναι το εξής. Εναπόκειται στον Πρόεδρο να προεδρεύει σε κάθε συζήτηση και όχι στα μέλη ε, της Επιτροπής, με κάθε σεβασμό πρέπει να σας πω, ότι έχω τον κατάλογο ομιλητών όλων των μελών που θέλουν να μιλήσουν και έχουμε προγραμματίσει χρόνο μέχρι τις 5.30 για τη συζήτηση αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τον κατάλογο των ομιλητών, βλέπω ότι προλαβαίνουμε ε, και μπορούμε να αφήσουμε και κανένα βουλευτή να ξεπεράσει το χρόνο του, όπως και εσείς κάνατε άλλωστε. Προσπαθώ να δείχνω όσο γίνεται περισσότερη κατανόηση. Δεν έχετε το λόγο κύριε Φέστη για να απαντάτε τώρα. Λοιπόν, ε, ο νοόν νοήτο. Καμιά φορά είναι πάρα πολλοί ομιλητέ και θα πρέπει να τηρούμε αυστηρά το χρόνο μας. Από την άλλη, μπορεί και κάποιος να υπερβεί το χρόνο που έχουμε προγραμματίσει, έτσι, μέσα σε λογικά πλαίσια, χωρίς να γίνει καμιά τρομερή ζημιά χρονική. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 5.30 για τη συζήτηση αυτή. Η κυρία Κανκό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ελπίζω παρόλη αυτή τη συζήτηση και μετά από όλα αυτά να παραμένει το δικό μου δίλεπτο. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα, κύριε Κίνγκ. Συνεργασία στα κράτη-μέλη για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκ των όνων κάνευ για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του εξτρεμισμού και για να υπάρχει ασφαλή ε, Ένωση. Ε, η ομάδα μου, η CR, ε, ήταν εμπνευστή ε, της νομοθεσία για το PNR και ήταν σημαντικό βήμα σε αυτή την αρχιτεκτονική. Ο Γιάνν Γιάνν Μπον, πρώην Βέλγος Υπουργό Εσωτερικών, πρωτοστάτησε σε όλα αυτά. Στη συνέχεια, το Βέλγιο ε, είδε να σημειώνονται επιτυχίες από το σύστημα αυτό. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα όμως για να εφαρμοστεί παντού στην Ευρώπη με τρόπο αποτελεσματικό. Όπως γνωρίζετε η εφαρμογή χωλαίνει, είναι μέγα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι το πιο συναρπαστικό θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, ποια είναι τα μαθήματα που μπορούμε να εξαγάγουμε από την ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού PNR εν ώψη οποιασδήποτε διεύρυνση σε αεροπλάνα, σε μάλλον σιδηρόδρομο και σε ε, πλοία. Είναι εξίσου προτεραιότητα για την έγκρισή του. Ευχαριστώ η κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι ε, θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ ικανός και πάρα πολύ δίκαιος όταν προεδρεύετε σε αντίθεση με κάποιον ομιλητή προηγουμένως. Εν ε, νομίζω ότι μιλήσατε για τους τζιχαντιστές, ξένους μαχητές, τρομοκράτες, ριζοσπαστικοποίηση. Κύριε Κίνγκ, θέλω να πω κάτι και λυπάμαι πάρα πολύ που τοσα πολλα πολλά κράτη-μέλη δεν το σκέφτηκαν αυτό όταν έδιναν όπλα στους και τους έστελαν στη Συρία σε ένα παράνομο πόλεμο ε, στο Ιράκ. Αυτές οι πράξεις έχουν και συνέπειες. Αυτό τους έκανε τρομοκράτες, εκεί που τους στείλαμε. Και καλά θα ήταν να σταματήσουμε να αναμειγνιόμαστε ε, σε τρίτες χώρες. Αυτό θα βοηθούσε πολύ περισσότερο την ασφάλεια ε, από την περιστολή των προσωπικών ελευθεριών και τον έλεγχο των συνόρων. Θέλω να επικεντρωθώ στα εξή δύο, κυρίως. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ασχολείται με τα θέματα ασφάλειας όταν τόσοι πολλοί υποψήφοι επιτροποί και οριστέντες ε, δεν έχουν χειριστεί σωστά ε, κάποια στοιχεία προσωπικά κτλ. Αναφέρομαι στον Σενιόρ ε, Ιωζέπ Μπορέλ που ξέρω ότι έχει διαδώσει προσωπικές διαβαθμισμένες πληροφορίες εμπιστευτικές στο Twitter ε, για την Ισπανία, ειδικά σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης πρώην ε, Υπουργού της Καταλωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ήταν εξωφρενική παραβίαση των κανόνων και των διαδικασιών. Και επίσης των αντίστοιχων ε, ε, οδηγιών ότι δεν μπορείς να βγάζεις τα social media και να δημοσιεύεις τέτοιες εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες. Γιατί, επειδή είναι καταλανή τα θύματα και δεν πειράζει, δεν μετράει, τι, η Ισπανία μπορεί να παραβιάζει τον νόμο. Η απάντηση της Ισπανίας ότι αυτό είναι ένα ενδοϊσπανικό θέμα. Δεν ισχύει αυτό, είναι ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Ο λόγο δεν θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχει πρόσβαση. Πόσο μάλλον να ε, το δημοσιεύει αυτό στα social media. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μάθω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγχει την πρόσβαση στην ίδια της τη βάση δεδομένων όταν παραβιάζονται τόσο κατάφορα οι κανόνες. Και δεύτερη ερώτηση ε, αφορά την εταιρεία του κυρίου Μπρετών, του Μεσχέ Μπρετών, και τι γίνεται με το ΣΥΣ, το, σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν. Και οι Βρετανοί θα ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους Αμερικανούς. Θα πρέπει ε, να μας ενημερώσετε εσείς και ο νέος Επίτροπος Βιομηχανίας δεν θα πρέπει να ενέχεται σε τέτοιες κατάφορες παραβιάσεις έτσι κι αλλιώς. Ε, λοιπόν, προτείνω τώρα, Επίτροπε, να απαντήσετε. Μάλλον όχι. Να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη, να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις και να απαντήσετε συνολικά στο τέλος. Η κυρία Μπρίκμο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Κίνγκ. Τα είπαμε τέλος Ιουλίου και ήδη είχαμε αναφερθεί στο θέμα επαναπατρισμού των παιδιών από τη Συρία και το Ιράκ και το μεταξύ κατάσταση άλλαξε πολύ. Αναφερθήκατε επίση και σε κάτι άλλο. Διευκρινίσατε ότι το, θέλουμε να το να μεγαλώνουν τα παιδιά σε τέτοια περιβάλλον με συγκρούσει είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι επιτόπιες εξελίξεις, τι άποψη έχετε από πάνω σε αυτό στην Επιτροπή Λίμπε την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε ενδιαφέρον το θέμα παρέβαση του κ. Βαντίφελ που είναι ο διευθυντή τη ΛΟΚΑΜ. Φορέα που ασχολείται με την ασφάλεια στο Βέλγιο και πραγματικά αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει κατεπηγούσα ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού. Όταν το συζητούμε αυτό σε πλαίσιο εθνικών κυβερνήσεων και στο Βέλγιο, οι υπουργοί μα λένε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι παίζουμε ένα πολιτικό πινκ-πονγκ εδώ. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν μετά τι τελευταίε μα συνομιλίε είχατε πιο στενέ επαφέ για καλύτερο συντονισμό με, στα πλαίσια του Συμβουλίου και με του συναδέλφου Τζόχανσον και Μπορέλ και τον Σαν Μισελ, τον μελλοντικό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που δήλωσε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα, κυρίως αφορά τις συζητήσεις για τις συγκρούσεις στα διάφορα μέρη του κόσμου. Το θέμα του επαναπατεσμού είπατε ότι δεν τίθεται πλέον μόνο για τα παιδιά, αλλά τίθεται και για θέματα ασφαλείας και για τους ενήλικες. Ποια είναι η απόψη σας επ' αυτού, διότι υπάρχει έλλειψη χρόνου για να δημιουργήσουμε ένα ad είναι πολύ κατεπήγον το θέμα. Καλύτερο να ελέγξουμε και να κρίνουμε αυτού τους ανθρώπους στα δικαστήριά μα παρά να τους αφήσουμε εκεί ελεύθερου. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ραγγέλ έχει το λόγο. Naturally, I want to praise your commitment. Σας επενώ για την προσπάθεια για διαφάνεια και λογοδοσία που αποδίδεται σε αυτό το κοινοβούλιο στον αφορά το σας. Σήμερα στο, στη Λίμπε από τον Ιούνιο, αλλά είναι σαφής υποχρέωση που έχετε αναλάβει και εφαρμόζεται. Σαν εισηγητής για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, σας διαβεβαιώ ότι έχουμε εργαστεί πάρα πολύ γρήγορα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ολοκληρώσει περίπου 15 ώρες διαπραγματεύσεων μετά τον πρώτο τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου. Ως εισηγητής και υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις εκ μέρου του Κοινοβουλίου, σας διαβεβαιώνω ότι κινούμεθα αρκετά γρήγορα από το τέλος Οκτωβρίου και μετά. Όμως, να υπογραμμίσω κάτι. Υπάρχει νομοθετικός λαβύρινθος ο οποίος ε, διερευνάται. Η νομοθεσία δεν είναι καλή κατά την άποψή μου. Έχουμε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τροποποιούν άλλες προτάσεις της ιδίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων και είναι τροποποιητικά κείμενα που έχουν εγκριθεί. Αυτό δεν βοηθά. Κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά τις διαπραγματεύσεις. Αυτό πιστεύω. Η διαδικασία δεν έχει εκπονήσει καλούς νόμους. Και αυτή η νομοθεσία δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατία. Το Κοινοβούλιο κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια αλλού παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει αυτοσυγκράτηση. Να μην αλλάζει προτάσεις που έχει υποβάλει και οι οποίες έχουν μάλιστα υποβληθεί αρκετά πρόσφατα. Τέλος. Να σχολιάσω δύο διαφορετικά θέματα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαστήκατε επί παραπληροφόρησης και επί ψευδών ειδήσεων. Πολύ καλή δουλειά. Το Κοινοβούλιο πρόσφατα τοποθετήθηκε είπε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, επενδύοντας περισσότερα. Ανησυχούμε διότι βλέπουμε ότι η οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών δεν έχει ενσωματωθεί μέχρι τώρα στο εθνικό δίκαιο των περισσότερων κρατών μελών συμπεριλαμβανομένη της, συμπεριλαμβανομένης πατρίδας μου της Πορτογαλίας. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση τωρινή, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Μπράιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την ε, παρουσίασή σας. Δεν θα σας εκπλήξει ότι διαφωνούμε ριζικά για τα μέτρα παρακολούθησης που επικαλείται η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, όπως η Οδηγία PNR η Ευρωπαϊκή, που είναι για μας παράνομη μαζική παρακολούθηση και σύμφωνα με την ομολογία του ε, ΔΕ και δεν θα σας εκπλήξει να ακούσετε ότι χρειάζεται πηγόντως μορατόριο για τη μαζική παρακολούθηση. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τον αντίστοιχο κανονισμό και το στείλατε στο Κοινοβούλιο για να συμφωνήσουμε, λέτε, κατεπηγόντω. Μπορούμε να συμφωνήσουμε και αύριο, αν υποστηρίξετε εσεί τη δική μας θέση και προσέγγιση και έκθεση. Πολύ, πολύ γρήγορα μπορεί να διεκπαιρεωθεί αυτό το θέμα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, αναφερθήκατε στην ασφάλεια του δικτύου 5G και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω τι πιστεύετε για την κρυπτογράφηση και από ε, κρυπτογράφηση. Ε, είναι σημαντικό αυτό γιατί οι κινέζικε εταιρείε ενέχονται βέβαια, αλλά και μπορεί οι επικοινωνίε να ε, ελέγχονται από μια τρίτη χώρα, από τι Πολιτείες. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Να κρυπτογραφούνται και ξέρετε και οι υπηρεσίε πληροφοριών και μυστικέ υπηρεσίε θέλουν και αυτέ να έχουν ασφαλή επικοινωνία. Και ένα τρίτο τελευταίο ε, και στην έκθεση και στην παρουσίασή σα. Αναφερθήκατε στην ε, αίσθηση του, κοινού για την ασφάλεια. Πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι η ζωή του είναι όλο και πιο επικίνδυνη, ότι αυξάνεται το έγκλημα, αυτά τα λένε τα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι συχνά ισχύει το αντίθετο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας, ε, ιδιαίτερα γιατί το εκμεταλλεύονται αυτό ε, ε, ακροδεξιοί, οι δεξιοί λαϊκιστές. Αυτό είναι και ει βάρο της δημοκρατίας, αν ο κόσμος νομίζει ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά του. Ενώ γεγονό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα ασφαλέστερα μέρη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Κίνγκ έχει περίπου 15 λεπτά για να απαντήσει. και να περάσουμε και στο τελευταίο σημείο που θα αφορά τα ηλεκτρονικά ε, αποδεικτικά στοιχεία. Ε, έχετε το λόγο κύριε Κίνγκ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους όσους ε, ε ασχολούνται με τα αισθήματα αυτά από όλες τις, ε, τις οπτικές γωνίες. Εμείς καλωσορίζουμε αυτές τις απόψεις, ε, τις συνεισφορές, ιδιαίτερα εάν θέλουμε να υπάρξει και μια θετική ανταπόκριση σε επίπεδο κοινή γνώμη. Συμφωνώ απόλυτα με το τελευταίο που υπόθηκε. Δεν θα συμφωνήσω για όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα, αλλά για το τελευταίο που είπατε, ε, πραγματικά πιστεύω ότι συλλογικά μα περιμένει μια πρόκληση. Πρέπει να διαχειριστούμε το πώ συζητούμε για τα ζητήματα αυτά και το τι κάνουμε για αυτά. Με έναν τρόπο που να ευαισθητοποιεί ε, τον κόσμο, χωρί όμω ε, να ε, δημιουργεί φόβο ή να ενισχύει το λαϊκισμό. Και δεν υπάρχει, δεν είναι, απλό, δεν είναι απλή απάντηση στο να βρεθεί λύση γι' αυτό. Πάντω δεν μπορούμε και να κρυβόμαστε από τα ζητήματα αυτά. Οπότε καλό είναι να γίνει αυτή η συζήτηση που ελπίζουμε να μας βοηθήσει όλους να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη σχέση και με, με την κοινή γνώμη. Για τα διάφορα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν με τη σειρά και εντάχει, αν ξεχάσω κάποιον, ε, θα επανέλθω. Για το επίπεδο των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τζιχαντιστική τρομοκρατία. Ακούστε, χωρίς ε, ε, να θέλω να είμαι, να είμαι ανησυχητικός, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος. Μετά το το θάνατο του Μπαγκδάτη, μια σειρά από χώρες ε, της Ευρώπης, μεταξύ των η Γαλλία έχουν ε, αλλάξει το επίπεδο συναγερμού, διότι θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνο. Σε κάποιε χώρε, μεταξύ των οποίων και το Ενωμένο Βασίλειο, έχουν χαμηλώσει το επίπεδο συναγερμού. Ε, δεν πάνε πάντα προ την ίδια όλα αυτά. Και αυτό είναι και μέρο τη γενικότερη ε, δημόσια συζήτηση. Ε, φοβάμαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ριζοσπαστικοποίηση. Ε, όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για εξτρεμιστές τζιχαριστές, αλλά και ακροδεξιούς ε, και άλλες μορφές ε, ε βίαιου εξτρεμισμού. Εμείς ε, εμένουμε και λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια λύση για το τρομοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά. Υπάρχει το θέμα της ρομαστικοποίηση της φυλακίας, βεβαίως και υπάρχει. Και πάλι, εδώ δεν θέλω να φανώ ανησυχητικός, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε γι' αυτό είναι περίπου 1.100 άτομα αυτή τη στιγμή ε, στις φυλακές ανά την Ευρώπη ε, που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, για τρομοκρατικές πράξεις. Αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν από τη φυλακή σε μερικά χρόνια. Ε, εκτιμούμε επίσης με βάση τις επιστροφές από τα κράτη-μέλη υπάρχει ένας ε, διπλάσιος αριθμός ανθρώπων που είναι στη φυλακή, που πήγαν στη φυλακή για άλλους λόγους αλλά που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, εκεί. Και αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση για μας. Για το πώς δηλαδή ε, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αντιμετώπιση όχι μόνο των ανθρώπων που βιώνουν τη φυλακή, αλλά και αυτούς που είναι στη φυλακή και που ριζοπαστικοποιούνται εκεί. Και έχουμε και το θέμα του ξένους μαχητές βεβαίως. Ε, τέθηκε ένα ερώτημα από τον κύριο Φέστ λέγει ότι δεν κάναμε τίποτα μετά τον Πατακλάν. Ε, δεν είναι έτσι. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μετά τον Πατακλάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συστηματική, συστηματικός έλεγχος εξωτερικά μας σύνορα. Έχουμε εξυγχρονίσει το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Υπάρχει υποχρέωση ε, συμφωνημένη να αλλάζουν πληροφορίε στα κράτη-μέλη για τα αισθήματα αυτά. Ε, δισεκατομμύρια φορέ ε, χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό με στοιχεία για ανθρώπου οι οποίοι έχουν ε, σχέση με τρομοκρατικέ πράξει. Έχουμε βελτιώσει την αλλαγή πληροφοριών, έχουμε βελτιώσει το σύστημα με το οποίο ε, συνεργάζονται η Europol και άλλα όργανα για να εντοπίσουμε ποιοι είναι επικίνδυνοι, ποιοι αποτελούν απειλή και προσπαθούμε αυτά ε, τα στοιχεία να τα έχουν οι υπηρεσίε, οι αστυνομικέ, οι τρομοκρατικέ, οι συνοριακέ. δεν είναι σωστό να λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ασφάλεια που εντοπίστηκαν πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, για την παραπληροφόρηση. Εδώ κάνουμε πολλά πράγματα. Αναφέρονται στην έκθεση, τα συζητήσαμε και την περασμένη φορά. Υπάρχει εδώ ε, η πρόκληση να μπορέσουν να συγκεντρωθούν τα κράτη-μέλη σε αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να είναι κάτι που θα ιδιωτικοποιηθεί και που θα το αναλάβουν κάποιες εταιρείες. Θέλουμε το αντίθετο. Γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια ε, στα πλαίσια των ευρωεκλογών να υπάρχουν, να υπάρχουν τα δίκτυα ε, ασφάλειας των εκλογών στα κράτη-μέλη, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για τις προειδοποίησει. Κάποιοι το επέκριναν αυτό, διότι ε, δεν ενεργοποιήθηκε, αλλά έκανε μια πολύ καλή δουλειά καθημερινά, δημιουργώντας ε, διασυνδέσεις με των κρατών μελών και των υπεύθυνων εκεί ε, για τα ζητήματα αυτά. Ε, θέλουμε να συνεργαστούμε βεβαίως με τον ιδιωτικό τομέα για τα θέματα αυτά, όχι όμως να ιδιωτικοποιήσουμε το έργο, τις αποφάσεις που θα παίρνονται. Αντιθέτως, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη διάδραση με ανεξάρτητους τρίτους ε, φορείς που θα παρακολουθούν τη διαδικασία και να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη διαδικασία ε, παρακολούθησης, ε, να υπάρχει σχετική πραγματογνωμοσύνη. Αυτή τη στιγμή αυτή η πραγματογνωμοσύνη ε, υπάρχει σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών, σε επίπεδο ερευνητών, σε επίπεδο ΜΚΟ. Ε, συμφωνώ μαζί σας όμως κυρία Σίπελ ότι αν δεν μπορέσουμε, μπορέσουμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο, πρόοδο πιο γρήγορα για τα ζητήματα αυτά Κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε, και αυτό θα το δει η Νέα Επιτροπή, είναι κατά πόσο χρειάζεται κάποιο άλλος διακανονισμό για την ανεξάρτητη αυτή ε, παρακολούθηση των δράσεων των κοινωνικών μέσων ε, στο ε, πολιτικό πεδίο, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ε. Γίνεται αυτό, να το αφήσουμε δηλαδή στα χέρια ε, εξαιρετικών κατά τα άλλα ε, εκπροσώπων ε, τη κοινωνία των πολιτών και ερευνητών ή είναι ένα ρόλο που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Τώρα, για τα ναρκωτικά. Δεν μιλάμε συχνά για τα ναρκωτικά ε, και θα έπρεπε, διότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση σε, σε ποινικό επίπεδο. Ε, ξέρετε τι κάνουμε για να μπορούμε να συντονιστούμε για τα ζητήματα των ναρκωτικών. Ε, τον ε, ρόλο της Europol, τον κύκλο ευρωπαϊκής πολιτικής. Τι προάλλες η Europol ανακοίνωσε ε, μια επιτυχή, κάποιες επιτυχές κοινέ ημέρες δράσης, επιτυχές κοινέ ημέρες δράσης ε, που έδωσαν έμφαση στο ζήτημα του ναρκωτικών και που οδήγησαν σε κατασχέσεις ρεκόρ σε συνθετικά ναρκωτικά. Αυτό δείχνει βέβαια ότι υπάρχουν και πιο πολλά συνθετικά ναρκωτικά αλλά και κατάσχεση 1.400 ε, κιλών ε, κοκαίνης και 110 συλλήψεις επίσης είχαμε συνολικά από αυτές τις επιχειρήσεις. Ε, εξακολουθεί λοιπόν να είναι σημαντική προτεραιότητα για μας. Τώρα για το PNR. Καλωσορίζω τη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα για το PNR. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα όπως θα θέλατε. Ε, θα συνεχιστεί όμως ο διάλογος αυτός και ενθαρρύνω, θα ενθαρρύνω τον ε, ε, διάδοχό μου να συνεχίσει το διάλογο αυτό, διότι έχουμε δουλειά. Θα πρέπει να κλείσει η συμφωνία με τον Καναδά και θέλουμε να το κάνουμε αυτό και συνεργαζόμαστε με όλους όσους ε, μπορούν να βοηθήσουν για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί κοινές, να ολοκληρωθούν οι κοινέ αξιολογήσει. ότι Εσεί ε, θεωρείτε ότι η διαδικασία των κοινών αξιολογήσεων δεν είναι ικανοποιητική. Εμεί όμω ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, η διαδικασία που συμφωνήσαμε όλοι, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που συμφωνήσαμε και εσεί βεβαίω θα, και εσά θα λογοδοτήσουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτέ οι αξιολογήσει θα είναι αποτελεσματικέ. Τώρα από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί και η συζήτηση για το PNR βεβαίω. Ε, και αυτό έχει να κάνουμε και με αυτό που είπε ο κ. Μπρίερ για την μαζική παρακολούθηση. Θα ήθελα απλώ να πω κάτι έτσι προσωπικά, χωρί να δεσμεύω κάποιον άλλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν θέλω να παρακολουθούμε μαζικά του ανθρώπου και δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό. Δεν έρχομαι εγώ εδώ για να παρουσιάσω, είναι περασπιστό οποιοδήποτε ευρωπαϊκό εργαλείο που διενεργεί μαζική παρακολούθηση Ευρωπαίων πολιτών. Και το PNR δεν το κάνει αυτό. Μπορεί να υπάρχει βεβαίως ε, μια ε, ουσιαστική διαφωνία εδώ. Τα, τα στοιχεία PNR συλλέγονται ούτω ή άλλω. Δεν κάναμε εμεί κάποιο εργαλείο για να τα συλλέγουμε. Ε, υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και πώς χρησιμοποιούνται. Ε, κάποια από τα στοιχεία λοιπόν που έχουν προκύψει για το πόσε πληροφορίες, αυτές τις πολλές πληροφορίες ε, όντω ε, εξετάζονται ή τα, τα τα ψάχνει κάποιος, διαπιστώσαμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία ε, των πολιτών των οποίων τα στοιχεία πιενάρα έχουν συλλεγεί δεν έχουν, εξετάζονται ποτέ. Δεν ενεργοποιούν κάποια τέτοια διαδικασία και αυτό είναι ε, καθυσυχαστικό. 99,96% των, των επιβατών ε, δεν εξετάζονται τα στοιχεία τους περαιτέρω. Δηλαδή 0,04% μόνο υπόκεινται σε περαιτέρω μελέτη και πολλές από τις υποθέσεις αυτές τελικά είναι απλά ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία, με το όνομα μάλλον. Ε, είναι πολλές περιπτώσεις λοιπόν, ε, είναι μάλλον ελάχιστες περιπτώσεις όπου ε, δίνεται συνέχεια. Και ορισμένε φορέ όμω φέρνει αποτελέσματα. Είχαμε μια έκθεση πρόσφατα από το Βέλγιο για τα αποτελέσματα που έχουν από την επεξεργασία δεδομένων PNR ε, από την βέλγικη μονάδα ε, πληροφοριών για επιβάτε ε, έω τον Αύγουστο φέτο. 331 θετικοί έλεγχοι, 4 άτομα σε περίπτωση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικά και επίσης ε, και κάποιες υποθέσεις απαγωγής παιδιών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αποτελεσματικά είναι τα συστήματα αυτά και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να μπορούμε να παρουσιάσουμε καλύτερα τα στοιχεία. Θα σας στείλουμε βεβαίως αμέσως ε, τα στοιχεία, την έκθεση αυτή. Ε, σίγουρα θα πρέπει πάντως να συνεχιστεί η συζήτηση. Είναι μια από τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να καθησυχάσουμε όχι μόνο εσά, αλλά και, το, και τους πολίτες. Δεν το κάνουμε αυτό ε, επειδή μας αρέσει. Ε, πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, ότι είναι νόμιμο και ότι είναι αναλογικό. Και αυτό σχετίζεται και με το ερώτημα αυτό για την ε, παρακράτηση δεδομένων για την οποία ρωτήσατε και αυτή η συζήτηση σίγουρα θα συνεχιστεί εγώ πιστεύω, το έχω ξαναπεί και το ξέρετε, μπορεί να συμφωνείτε ή όχι, ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και η παρακράτηση των δεδομένων αυτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την επιβολή του νόμου και συνεισφέρει στην ασφάλεια των πολιτών μας. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνεται με έναν τρόπο που θα υπάρχει πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλαμβάνουμε εμείς και αποτυπώνεται και στην απόφαση του δικαστηρίου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα κάποιων υποθέσεων που εκκρεμούν. Παράλληλα ε, εργαζόμαστε για να βρεθούν κάποιες λύσεις, διότι δεν συμφωνούν όλοι για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Και εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε να το κάνουμε αυτό σε πλήρη διαφάνεια ε, απέναντί σας. Τώρα για τον για την πρόκληση των ξένων μαχητών, όχι τον κίνδυνο, τον πρόκληση ε, που ανέφεραν δύο βουλευτές εδώ, τι κάνουμε για ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή αυτή ε, και θέλουν να επιστρέψουν, έχουν ζητήσει να επαναπατριθούν Ακούστε, όπως και οι δύο είπατε πολύ σωστά, η νομική κατάσταση είναι η εξή, είτε μας αρέσει είτε όχι είναι ένα θέμα ευθύνης των κρατών μελών. Και βεβαίως αυτό το, ε, το, την αρμοδιότητα δεν την μοιράζονται τα κράτη-μέλη. Θέλω να προωθήσουμε εμείς μια συζήτηση για την κλίμακα και τη φύση του προβλήματος ε, για να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε μεγαλύτερο συντονισμό για τα ζητήματα αυτά. Εγώ ε, δεν το έχω θέσει απευθεία με τον Σαλ Μισελ, το έχω θέσει με άλλα του, σε άλλα μέλη του Συμβουλίου. Είχαμε μια συζήτηση από την τελευταία φορά στα πλαίσια της ομάδας G16 όπου εδώ καλύπτουμε και τους ενήλικες και τα παιδιά. Ε, εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησαμε να μοιραστούμε και να δημοσιοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία για την κλίμακα της πρόκλησης αυτής. Έχω δημοσιοποιήσει μια σειρά από στοιχεία για τον αριθμό των ενηλίκων που θεωρούμε ότι ε, βρίσκονται στην περιοχή αυτή, ε, ενήλικους που θεωρούμε ότι κρατούνται αυτή τη στιγμή, περίπου 600 άτομα και βεβαίως υπάρχει μια επιπλέον πρόκληση μιας και κάποιοι ενήλικες ε, βρίσκονται πλέον ε, υποκράτηση στην Τουρκία και οι Τούρκοι είπαν ότι θα έρθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης προσπάθησα να δημοσιοποιήσω τους αριθμούς που αφορούν στα παιδιά, διότι συμφωνώ και με τους δυο σα ε, το ζήτημα του τι θα κάνουμε με τα παιδιά επίγει. Υπάρχουν περίπου 1.400 παιδιά στην περιοχή που εμείς θεωρούμε ότι έχουν έναν γονέα ή και τους δύο Εκεί ε, ε, είναι υποκράτηση, η μισή από αυτού εκεί, κάποιοι άλλοι είναι σε στρατόπεδα. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά αυτά, διότι ο επαναπατρισμό των παιδιών επίση δημιουργεί πολλά ζητήματα. Αυτό φάνηκε και με την εμπειρία των κρατών μελών που επαναπάτρισαν κάποια παιδιά, ιδιαίτερα ορφανά. Πολλά παιδιά όμως που είναι κάτω των 6 ετών ε, να τα αφήνουμε στο έλεος ε, πολλών και διάφορων ε, καταστάσεων δημιουργούν πολλά ζητήματα ανθρωπιστικά αλλά και προκρόθεσμα και ζητήματα ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τα κράτη-μέλη να εξετάζουν το θέμα αυτό επιγόντως. Μιας και μιλάω για παιδιά, ε, μιλήσατε για την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών ε, και τα στοιχεία για την πραγματική εφαρμογή ε, ίσως έχετε δίκιο που το αναφέρετε ε, έχουμε μια ε, κακή εφαρμογή από 23 κράτη-μέλη. Δεν, δεν σημαίνει μέσα ότι δεν κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη. Ε, γίνεται μια προσπάθεια να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να έχουμε μια αποτελεσματική εφαρμογή. Και εξακολουθούμε να θέτουμε στα κράτη-μέλη αυτά μια σειρά αποζητήματα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και αυτό με φέρνει τώρα με οδηγεί στο ερώτημα της κυρίας Ντέλη για διάφορες πτυχές της χρήσης του ΣΥΣ, του Συστήματος Πληροφοριών Σέγγεν. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε πολλούς άλλους, παίρνουμε πολύ σοβαρά το θέμα της πραγματικής εφαρμογής, της πραγματικής χρήσης των ε, εργαλείων αυτών. Το σύστημα ΣΥΣ είναι σαφέστατο στο ποια είναι η χρησιμότητά του. Είναι ένα ε, σύστημα για την ε, εμπιστευτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και θα λογοδοτούν τα κράτη-μέλη για μια σωστή εφαρμογή του συστήματος αυτού. Όμως και εδώ, εδώ και άλλη μια φορά οι κανόνες είναι σαφείς, είτε συμφωνείτε είτε όχι. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν ποια είναι η αρμόδια αρχή, και ποιο έχει πρόσβαση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι αυτά στα οποία πρέπει να απευθύνει κανείς οποιαδήποτε ερώτημα για τη χρήση του ΣΥΣ. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουμε να κάνουμε αξιολογήσεις ε, Σέγγεν. Έχουμε το σύστημα ΣΕΒΑΛ, όπου έχουμε διάλογο με το καθένα από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν για το πώ χρησιμοποιούν το ΣΥΣ. Και θα συνεχίζουμε να ε, εκπονούμε εκθέσεις γι' αυτό και θα σας τις ε, δείχνουμε. Όχι ανοιχτά βέβαια, αλλά μπορείτε να έχετε εμπιστευτικά πρόσβαση ε, για να διαβάσετε αυτές τις εκθέσεις. Και μπορούμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό, να το συζητήσουμε με τη γραμματεία. Και με, στην προηγούμενη θητεία συνεργαστήκαμε με μια ομάδα από εσά που εξέταζε το πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΣΥΣ. Και αν το, αυτό το νέο κοινοβούλιο θέλει να δημιουργήσει μια αντίστοιχη διαδικασία εδώ με την γραμματεία, εμεί ευχαρίστω να την συνεχίσουμε. Και φαντάζομαι ότι και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει αντίρρηση. Μπορείτε να θέσετε εκεί λεπτομερή ερωτήματα. Τέθηκε ένα ερώτημα για τι δραστηριότητε μια ιδιωτική εταιρεία. Θα ήθελα εδώ απλώ να πω, χωρί να μπω σε λεπτομέρειε, διότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ δημόσια, ότι δεν απαγορεύεται από του κανόνε να χρησιμοποιήσει κάποιος μια ιδιωτική εταιρεία ε, για ε, υπηρεσίες ε, πληροφορικής και για συντήρηση συστημάτων. Δεν είναι το ίδιο με την πρόσβαση στι πληροφορίες. Τέλος, για το άλλο ερώτημα του, της κυρίας Μπρίες, θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ότι αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά. θα να υπάρξει πρόοδο είναι κάτι που συζητείται στους τρίλογου. Ε, ο τρίλογο είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευση. Ε, σε αυτόν τον τριμερή διάλογο λοιπόν, ε, εγώ δεν θα επιμείνω να παραμείνει κάθε γραμμή του αρχικού κειμένου τη Κομισιόν. Ελπίζω όμω και τα άλλα θεσμικά οργάνα και το Κοινοβούλιο δηλαδή και το, το Συμβούλιο να μην επιμείνουν ε, να τηρηθούν κατά γράμμα οι θέσει του για να σημειωθεί και πρόοδο. Διότι αυτό είναι και το πνεύμα ε, μια τέτοια διαδικασία του τριλόγου. Τώρα για την κρυπτογράφηση. Εγώ υποστηρίζω την κρυπτογράφηση. Το έχω πει αυτό πολλέ φορέ. Δεν θα ήθελα ο τραπεζικό λογαριασμό να μην είναι κρυπτογραφημένο. Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως με το 5G και με άλλες νέες τεχνολογίες, τις οποίες γνωρίζετε, ε, είναι πώς θα προφυλαχθούμε από την πρόσβαση σε πληροφορίες ε, σε άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να έχουμε και έναν διακονονισμό που να είναι αποτελεσματικό ε, για να έχει κάποιο πρόσβαση κατόπιν άδεια, ιδιαίτερα σε, από αρχέ υποβολή του νόμου, στα πλαίσια μια ε, δικαστική διαδικασία. Και αυτό είναι πρόκληση. Είναι μια διαφορετική τεχνική πρόκληση, ανάλογα με το για ποια τεχνική τεχνολογία μιλάμε. Η κρυπτογράφηση σχετίζεται με πολλέ και διάφορε τεχνολογίε. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Πρέπει να συνεχιστεί, Θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση χωρί άδεια ε, στα στοιχεία αυτά, χωρί όμω να κλείνουμε ε, το δρόμο στο να έχει κάποιο τελικά πρόσβαση κατόπιν άδεια βέβαια. Αυτά Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να έρθω. Ελπίζω ε, να ολοκλήρωσα έγκυρα την μου. Ακριβώς την ώρα μας. Γιατί έχουμε κι άλλο ένα θέμα και πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Και αυτό συνδέεται με την ασφάλεια όπως και η δικαστική συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου. Ε, σίγουρα όλα αυτά και ανεξαρτήτως της σύνθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φοντερ Λάιεν και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο που να επιγράφεται θέματα ασφαλείας, αυτά τα θέματα χρειάζονται συζήτηση σε βάθος εδώ στην Επιτροπή μας, γιατί μας ανησυχούν και μας αφορούν. Και όλες αυτές οι προκλήσεις στις οποίες αναφερθήκατε εσείς έχουν να κάνουν με το πώς θα συνδυάσουμε τώρα τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ε, δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή με ασφαλιστικές δικλείδες και χέγγια απέναντι στην τεχνολογική επανάσταση που ζούμε εδώ και κάποια χρόνια τώρα. Αυτή είναι η πρόκληση και θα παραμείνει και αναμένεται μια σωστή νομική απάντηση από τον Ευρωπαίο νομοθέτη αλλά από εμάς ακριβώς, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε για την προθυμία που δείχνετε πάντα να έρχεστε και να συζητάτε μαζί μας όσο μπορείτε. Now, no Λοιπόν, δεν κάνουμε διαλύματα τώρα και διακοπές, προχωρούμε. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολή και Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρηση Ηλεκτρονικών Αποδεικτικών Στοιχείων σε ποινικέ υποθέσει. Σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα το πλαίσιο. Είχαμε πρώτα μια πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το θέμα αυτό που σας ανέφερα. Στη συνέχεια έχουμε δεύτερη πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εναρμονισμένους κανόνες για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Όλο αυτό θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο νομικό για να συλλέγονται ηλεκτρονικά στοιχεία δεδομένα, αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου. Όταν υπάρχει υποψία διάπραξης αξιόπινης πράξης και δεν είναι ε, ούτε κατασταλτικό μέτρο, ούτε αστυνομικό, ούτε πρόληψης. Υπάρχει επίση το θέμα του ορισμού των νόμιμων εκπροσώπων στους παρόχους υπηρεσιών ε, ε, ιδιαίτερα όσοι παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουν ένα νόμιμο εκπρόσωπο. Το Δεκέμβριο του 2018 ενέκρινε μια απόφαση το Συμβούλιο, ωστόσο οκτώ υπουργοί προηγουμένως σε επιστολή τους εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξύντλησε τη συζήτηση στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο με διαβουλεύσεις με ενεχομένου, ενδιαφερομένους, δικαστικούς, εισαγγελεί. Ε, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πανεπιστημιακούς και δημόσια κρούαση ακόμα κάναμε και μια σειρά εγγράφων είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας από το Δεκέμβριο του 18 μέχρι τον Απρίλιο του 19. Γνωρίζετε ότι ετέθηκαν πολλά, πολλά νομικά ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, τις κατηγορίες δεδομένων, της αρχής ε, αναλογικότητας, ε, τις δυνατότητες προσφυγής. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε μια νέα ερμηνεία του άρθρου 82 τώρα, που είναι η νομική βάση. Ε, από την ε, Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν είναι, λέει, ακριβώς ποινικό δίκαιο. Και ούτε ακριβώς η δικαστική ποινική συνεργασία που είχαμε στο μυαλό μας. και έχουν να κάνουν με τις επαφές μιας διοκτικής αρχής σε ένα κράτος μέλος με ένα πάροχο υπηρεσιών ε, σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να υπάρχει πρώτερη ενημέρωση ούτε δυνατότητα αντίδρασης των εν λόγω διοκτικών αρχών στη δεύτερη χώρα. Είναι κάπως προβληματικό αυτό και μπορεί να τίθεται εδώ θέμα ετεροδικίας. Και θα έχουν ιδιωτικοί φορείς ε, νομικό ρόλο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό μας απασχόλησε τόσο πολύ καιρό αυτό το θέμα. Και τώρα ερχόμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Το 5 και το 6. E. Το ένα αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή για τη, τα, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Είναι κανονισμός και το άλλο είναι οδηγία για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων. Ας ακούσουμε την εισηγήτριά μας πρώτα, την κυρία Σίπελ, και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις με πρώτους τους συντονιστές. Έχετε το λόγο κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ελπίζω και οι σκιώδες να έχουν κάτι να πούνε ε, σε αυτό το γύρο της συζήτησης που θα κάνουμε. Ας αρχίσω απλούστατα με μία δήλωση επανερχόμενη στη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και συζητούσαμε τη Διεθνή Συμφωνία για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Και πάλι δείξαμε πόσο άρρηκτα συνδεδεμένα είναι τα δύο θέματα. Με μεγάλη μου απογοήτευση άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Χαίρομαι που δεν θα ολοκληρωθεί τίποτα ε, πριν ε, περάσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά, αλλά στο μεταξύ διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς ε, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ποτέ μια επιτροπή της Κομισιόν, ούτε στην επιτροπή μας, ούτε πουθενά, δεν βγαίνει ως τελικό προϊόν με την ίδια μορφή με την οποία κατατέθηκε η εντύπωση που έχω εγώ τουλάχιστον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προεξοφλήσει, να δημιουργήσει τα τελεσμένα ε, σε ό,τι αφορά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Τούτων λεχθέντων, Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι ε, για τη συνεργασία του σκιώδη ηγητές. Πρέπει να σας πω ότι ελέγξαμε σε μεγάλο βάθος την πρόταση αυτή, η οποία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια τελείως νέα προσέγγιση. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου, από τότε που έκανε την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς ως Επιτροπή Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ και ιδιαίτερα μαζί με τους σκιώδεις συναδέλφους, ε, Εργαστήκαμε πάρα πολύ επί των προτάσεων αυτών. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις και των σκιωδών και διμερείς, ακρόαση στην Επιτροπή μας και επτά έγγραφα εργασίας ε, βάσει όλων αυτών έρχομαι να σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο έκθεσης. Τι θέλω να σας προτείνω. Όπως βλέπετε στο σχέδιο έκθεσης, στα δύο σχέδια, προτείνω να απορρίψουμε την πρόταση οδηγίας και να εντάξουμε τα σημαντικά τμήματα της οδηγίας αυτής στον κανονισμό και να έρθουμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό με 267 συνολικά τροπολογίες. Για ποιο λόγο να απορρίψουμε την πρόταση οδηγίας. Απλούστατο. Για λόγους νομικής και πρακτικής συνέπειας. Η οδηγία που προτείνεται βασίζεται στο άρθρο 53 και στο άρθρο 62 της συνθήκης που έχει να κάνει με την αναγνώριση των πτυχίων και άλλων ε, τυπικών προσόντων και συντονισμό ε, για ε, υπηρεσίες, δράση διοικητική κτλ. Αυτή η οδηγία δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι ε, ότι ο κανονισμός θα δεσμεύσει μόνο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στα νομικά εργαλεία ε, που εγκρίθηκαν με βάση το άρθρο 4 κεφάλαιο 4 της συνθήκης. Άρα έχουμε μια δυσαρμονία, γιατί ο κανονισμός δεσμεύει μόνο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν, ενώ μια οδηγία ε, θα ε, δέσμευε με όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα πρέπει να ορίσουν νομικό εκπρόσωπο με βάση την οδηγία χωρίς να συμμετέχουν στον κανονισμό ε, για ε, τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Επιπλέον, με την οδηγία Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εισαγάγει την ιδέα του νομικού εκπροσώπου όχι μόνο για τα θέματα ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και για μελλοντικά ε, ε, μέσα για την αμοιβαία αναγνώριση. Και με ένα σαφή μηχανισμό κεντρικό συντονισμού που δεν εντάσσεται ούτε ε, στον κανονισμό ούτε στην αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης. Θυμίζω ότι η προστιθέμενη αξία της αμοιβαία αναγνώρισης ήταν ότι εισήγαγε άμεση επαφή μεταξύ των δικαστικών αρχών και ε, όχι των κεντρικών διοικητικών αρχών. Λυπάμαι, αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εδώ το έχετε παρακάνει και παρερμηνεύετε τη νομική βάση ε, της οδηγίας στο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες. Εγώ πιστεύω ότι μόνο τα κρατη που συμμετέχουν στον κανονισμό θα πρέπει να δεσμεύονται από οποιαδήποτε υποχρέωση σε ό,τι αφορά ε, τον ορισμό ε, ενός εκπροσώπου ο, ε, για την παροχή υπηρεσιών, ε, για την ε, εντολή υποβολής και Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρησης. Το άρθρο 53 δεν είναι υγιής νομική βάση. Γι' αυτό προτείνουμε τα στοιχεία αυτά να φύγουν από την οδηγία και να μπουν στον κανονισμό. Υπάρχει δυνατότητα αυτή με βάση το άρθρο 82 ως συνοδευτικό μέτρο. Το τσεκάραμε αυτό νομικά, τουλάχιστον εγώ το κοίταξα. Ε, οι πάροχοι τρίτων χωρών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν στο μέτρο είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν νομικό εκπρόσωπο. Αυτή η έννοια του νομικού εκπροσώπου για παρόχους τρίτων χωρών δεν είναι καινούρια, αλλά αντανακλά ας πούμε το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ε, GDPR. Ε. Αυτά όλα είναι πιο αποτελεσματικά και πιο συνεκτικά. Τι άλλο έχουμε. Α, διαδικασία κοινοποίηση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, επιτρέπει στις αρχές ε, που εκδίδουν την εντολή να απευθύνονται στους παρόχους χωρίς αυτόματα να απευθύνονται στις κρατικές αρχές όπου εδρεύει ο πάροχος. Αυτό είναι μια τελείως καινοφανή ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση σε ποινικέ υποθέσεις. Και αυτό επικρίνεται όχι μόνο από ειδικού σε ΜΚΟ για θέματα προστασίας ε, δεδομένων, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άλλους. Ακόμα και 8 κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ξέφρασαν έντονες επικρίσεις ε, σε μια επιστολή τους στην Προεδρία. Τους έλειπε ένα κράτος μέλος μόνο για να μπροκάρουν την απόφαση. Αυτό γιατί δεν πρέπει μας να μας απασχολεί. Φανταστείτε, εάν ένας πάροχος στο δικό μου κράτος μέλος υποχρεούται άμεσα από μια τρίτη διοκτική αρχή να ε, διατηρήσει ή να αποκαλύψει δικά μου προσωπικά δεδομένα χωρίς να το γνωρίζει αυτό το κράτος μου. Το κράτος μου αμελεί την ε, βασική του υποχρέωση να εγγυάται το σεβασμό των δικών μου θεμελιωδών κομμάτων στην επικράτειά του. Ε, δεν ευσταθεί νομικά η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δικαστή ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είπε και παραθέτω και τα 28 κράτη-μέλη και ε, τα υπόλοιπα που είναι συμβαλόμενα στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούνται να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επικράτειά τους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δημιουργεί μια μοναδική μάλλον κατάσταση σε σχέση ε, με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, συνεχίζει ο δικαστής. Ενδεχομένως ε, υπάρχει θεμητή προσδοκία ο νόμος της λόγω χώρας να εφαρμόζεται παντού. Και αυτό αντανακλά το σύνομο αυτής της πρότασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν απάντησε σε αυτή την επίκριση. Έχουμε μεγάλες διαφορές ε, στην ποινική ε, νομοθεσία που παραμένει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αρνηθούν ε, αυτές τις προτάσεις βάσει του νέου άρθρου 11α. Όλα αυτά συνάδουν σε όσα είχαμε ε, αποφασίσει για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας και δευκολύνει πολύ τη ζωή των επαγγελματιών του κλάδου. Ε, μια κοινοποίηση με νόημα και δικαίωμα αντίρρησης της ε, εκτελεστικής αρχής θα βοηθήσει πολύ και τους παρόχους των υπηρεσιών. Χωρίς μια τέτοια κοινοποίηση, οι ελεκτές των δεδομένων δεν μπορούν να είναι βέβαιοι αν γίνεται σεβαστή η νομοθεσία των κρατών στα οποία εδρεύουν. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανονικά θα πρέπει να αναθέτει σε εκείνου και όχι σε εταιρείε, αν οι εντολέ ε, είναι σύνομε ή όχι. Ε, νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Συνεπώ, προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολή και η Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρησης να αποστέλλονται ταυτόχρονα στο πάροχο υπηρεσιών και στην εκτελεστική αρχή. Απουσία οποιασδήποτε αντίρρηση τη εκτελεστικής αρχής σε ένα δεδομένο ορισμένο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένος ο πάροχος υπηρεσιών να υποβάλει ή να διατηρείται ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία ή να τα ε, ε, αποκαλύπτει στην ε, εκδούσα αρχή σε περίπτωση που το λόγο πρόσωπο δεν είναι ούτε πολίτης ούτε διαμένων στη συγκεκριμένη χώρα, μπορεί να φαίνεται αυτό περίεργο ή σπάνιο, ε, ε, αν είναι αυτό σαφές τη στιγμή της έκδοσης Ευρωπαϊκής Εντολής, ότι δεν είναι ούτε κάτοικος ούτε πολίτης της Ένωσης ε, στο κράτος που εκδίδει εκτελεί, θα πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνεται το κράτος διαμονής του. οι εντολές υποβολής είναι πιο ε, επιθετικές εντός εισαγωγικών ως προς τα προσωπικά δεδομένα από τις εντολές διατήρησης. Ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τα, ε, τις ασυλίες και ε, τα προνόμια, ε, αυτό είναι ένα θέμα του κράτους που όπου διαμένει μόνιμα ο ενδιαφερόμενους. Και μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται αυτή η κοινοποίηση να επί, ε, βραδύνει τις διαδικασίες. Είναι ένα δεκαήμερο. Ε, είναι το ίδιο διάστημα που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ωστόσο, θα πρέπει για τις επίγουσε περιπτώσεις να διευρυνθεί η προθεσμία να παραταθεί, ιδιαίτερα όταν είναι μικρή η υπηρεσιών και ε, έχουν περιορισμένους πόρους ανθρώπινους και τεχνικούς. Ε, θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές οι προθεσμίες και φυκτές. Ε, παρατείνοντας τις προθεσμίες από 6 σε 24 ώρες για τις κατεπήγουσες περιπτώσεις, είμαστε βέβαιοι ότι έχουν μια ολόκληρη εργάσιμη μέρα, μάλλον ολόκληρη μέρα, να ελέγξουν τα δεδομένα ε, ε, και το σύνομο ε, χωρίς να επιβραδύνεται πολύ η διαδικασία. Τι γίνεται με τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων προσώπων, των θυγόμενων. Ορισμένες από τις τροπολογίες μου τα καλύπτουν αυτά τα δικαιώματα και έχουν στόχο να ευθυγραμμίσουν τον προτινόμενο κανονισμό με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση και τη διεθνή νομοθεσία και την ομολογία. Μερικά παραδείγματα το να αυξηθεί το κατόφλι για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής από τρία χρόνια σε πέντε χρόνια κάθερξη. Αλλιώ τα κράτη-μέλη, σε πολλά κράτη-μέλη, φτάνουν όλα τα κακοργήματα και τα μικρά εγκλήματα στην τριετή φυλάκιση. Υπάρχει ένας κατάλογος 32 κακουργημάτων που θεωρούνται σοβαρά εγκλήματα σε ε, όλα τα προηγούμενα μέσα αμοιβαία αναγνώρισης και μεταξύ αυτών ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Επανέρχομαι στην ε, σαφή διάκριση του περιεχομένου Σύμφωνα με την ε, νομοθεσία, ε, και η διακίνησή τους και η ε, διατήρησή τους χρειάζονται εγγυήσεις όχι μόνο στην έκδοση αλλά και στην εκτέλεση των εντολών υποβολής και διατήρησης. Υπάρχει θέμα του απαραδέκτου στο δικαστήριο της ε, διαγραφής δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα κλπ. Επίσης υπάρχει ένα θέμα ορολογίας, ηλεκτρονική ενημέρωση, electronic information. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι είναι παραδεκτά ως ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία στις ποινικέ υποθέσεις. Αυτό όμως δεν ισχύει κατά ανάγκη. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση μπορεί να αντικατασταθεί ε, ε, και αυτό δεν προεξοφλεί ή δεν προεξοφλούμε εμείς την αξία των δεδομένων. Ε, είναι ρόλος του δικαστηρίου στη διαδικασία να αξιολογήσει αν είναι παραδεκτά αυτά τα στοιχεία ή όχι. Τελευταίο θέμα, σύγκρουση νομοθεσίας με μια τρίτη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια ειδική επιτροπολογία σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση με τρίτα κράτη και αφήνει ε, την τελευταία απόφαση στην εκδούσα αρχή και σε μερικές περιπτώσεις ε, τις αρχές ε, της τρίτης χώρας. Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία δεν προβλέπει προθεσμίες καθόλου. Και τι θα γίνει τώρα, θα είναι μια τέρμονη ιστορία αυτή. Αντί να αφήνει την τελική απόφαση στην εκδούσα αρχή, θα πρέπει η εκτελεστική αρχή, ε, ε, να, η εκτελούσα αρχή να αποφασίσει, ε, γιατί στο δική της επικράτεια τελείται το, η παράνομη πράξη, η αξιόπινη. Τελικό συμπέρασμα. Το βασικό επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν και παραμένει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Όταν ενέκρινε ε, λίγους μήνες αργότερα την απόφασή της, το Συμβούλιο, ε, το βασικό επιχείρημα ήταν και παραμένει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των περισσότερων χωρών. Ε, αναγνωρίζω τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν σήμερα οι διοκτικές αρχές αλλά η αποτελεσματικότητα ευσταθεί ως επιχείρημα εάν ταυτόχρονα ε, υπάρχουν τα εχέγγυα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία ε, των ελευθεριών. Οι τροπολογίες που προτείνω θα εξασφαλίσουν ε, να δημιουργήσουμε ένα νομικά υγιές και αποτελεσματικό νομικό εργαλείο που θα αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα, θα δίνει ασφάλεια δικαίου για τις αρχές, τους παρόγους υπηρεσιών και τους θυγωμένους ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας απολύτως το σεβασμό των ανθρωπίνων ε, και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ και πάλι τους κιόδης και περιμένω να ακούσω τους υπολείπους. Ευχαριστώ. Okay, as the two previous points... Ευχαριστώ. Στο γύρο των συντονιστών, λάθος είπα συντονιστές. Τους κιόδης ε, πρέπει να αναφέρω. Ο κύριος Βέντοχο από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Λέω ο κύριος Μέλο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια. Έκανε πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα και μας έκανε και προτάσεις. Περιπλοκότατο ζήτημα, δυσχερέστατο και δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν όλοι πάνω σε αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι έκανε πολύ δουλειά. Έκανε πάρα πολύ δουλειά. Ας δούμε ποιος ήταν ο στόχος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Χρειαζόμαστε ψηφιακή συνεργασία και σχετικούς μηχανισμούς. Να είμαστε έτοιμοι για την ψηφιακή εποχή, για τη συλλογή στοιχείων διότι πολλά εγκλήματα είναι έξω από την εμβέλεια στην οποία μπορεί να κινηθεί η δικαιοσύνη. Είναι πολύ τεχνική η φύση του θέματος, χωρίς σύνορα, όμως πρέπει να αποδίδεται αποτελεσματική δικαιοσύνη. Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί για την παραγωγή και διατήρηση στοιχείων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ. Δεν υπάρχει ταχεία μέθοδος για να γίνει αυτό. Και αυτοί που ουσιαστικά ωφελούνται είναι οι εγκληματίες. Πρέπει να διαφυλάσσουμε τα ατομικά δικαιώματα, κυρίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Δεν πρέπει να κρύβουμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα των οικονομικών εγκλημάτων που προσπαθούμε να καλύψουμε, παρόλο που είναι σημαντικό τομέα, αλλά μιλάμε για όλες τις μορφές ε, εγκλημάτων χωρίς σύνορα είναι εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας, όπου οι εγκληματίες πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από τις εισαγγελικές αρχές. Βασίζονται στην έλλειψη συνεργασίας, ούτως ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται στις παράνομες δραστηριότητές τους. Και χρειάζεται να είναι ισορροπημένη η ανταπόκρισή μας, να εξασφαλίζουμε ότι πραγματικά αποδίδεται δικαιοσύνη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πλήρης προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι πολύ ευμετάβλητα αυτά τα στοιχεία, αυτού του είδους τα στοιχεία. Δεν πλαισιώνονται από σύνορα και δεν μπορούν να μεταδίδονται από παραδοσιακές διάβλους. Εδώ και κάποια χρόνια ήμουν εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Αυτό το ένταλμα έρευνας είναι ένα πρόσφατο εργαλείο, αλλά δεν κάλυπτε αυτού του είδους τα στοιχεία που συζητάμε τώρα. Οι διαπραγματεύσεις και τότε ήταν πολύ δύσκολες. Γι' αυτό αυτά τα, θύμα, τα θέματα δεν είχαν καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Υπάρχει η ανάγκη οι δικαστικές αρχές να έχουν τους αναγκαίους πόρους. Χρειάζεται όμως να διεξάγονται οι αναγκαίοι δικαστικοί και συνταγματικοί έλεγχοι στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται μια σωστή ισορροπία. Διαφωνώ με κάποιες προτάσεις ηγήτριας. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Ιδεοδός θα έπρεπε να βρούμε κάποια συνένεση. Πρώτα απ' όλα διαδικασία κοινοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Αλλά να μην υπάρχει κανένα δικαστικό έλεγχο από το κάτω μέλο. Το κάτω μέλο απαραίτητα από αυτό. Στι 30 Νοεμβρίου προτάθηκε αυτό στο Συμβούλιο είπε να προβλέπεται μια διαδικασία κοινοποίηση για δεδομένα που αφορούν περιεχόμενο. Οι πάροχοι ε, των υπηρεσιών που είναι ιδιωτικοί φορεί, θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους νομιμότητας αλλά δεν είναι δικαιοδοτικά όργανα. δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτοί οι φορεί αποφάσει, πρέπει να είναι αποφάσει του δικαστικού κλάδου. Και αυτό το σύστημα κοινοποίησεω ξεπερνά τα όρια του αναγκαίου. Είναι περιπλοκότατο και δεν θα είναι παρακόρως αποτελεσματικό. Ενώ για αυτό του είδου τα προβλήματα, τα εγκλήματα πρέπει να έχουμε ταχύτατο σύστημα, αποτελεσματικότατο. Πολλέ προτάσει θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα δεν θέλουμε να περιπλέξουμε το μέσο παραπάνω από ό,τι πρέπει, να είναι πιο περίπλοκο από το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνα. Το αντίθετο πρέπει να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση που κουβεντιάζουμε. Να δώσω και κάποια παραδείγματα. Καθορισμός διαφόρων κατηγοριών δεδομένων. Αυτή είναι μια νέα ιδέα της εισηγήτριας. Προ, ε, δεδομένα για την πρόσβαση και δεδομένα για τις συναλλαγές και ε, γραφικά στοιχεία είναι μια νέα κατηγορία, εικόνες, απεικόνηση. Ε, πώς όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στα διάφορα ποινικά συστήματα. Νομίζω ότι έτσι η πρόταση γίνεται λιγότερο ε, αποτελεσματική. Δεδομένα για την πρόσβαση, access data, χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη. Γι' αυτό το λόγο και μόνο χρησιμοποιούνται. δεν είναι τόσο δυσδυτικά, παρεμβατικά όπως τα δεδομένα που αφορούν συναλλαγές που επιτρέπουν τη δημιουργία μιας εικόνας, μιας φωτογραφίας, μιας απεικόνησης του χρήστη. Αν συνδυαστούν αυτά με τα δεδομένα περί προσβάσεων, τότε δημιουργείται μια νέα κατηγορία και σε πολλές περιπτώσεις οι ερευνητικές αρχές δεν θα είναι σε θέση να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τον εικαζόμενο εγκληματία που είναι το πρώτο στο βήμα στην έρευνα. Άρα περιπλέκουμε το έργο τους. Ευθύς εξ αρχής, όταν προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τον υπεύθυνο για το έγκλημα. Μετά, νέο ορισμό για τα δεδομένα τα σχετικά με το περιεχόμενο. Αυτή είναι μια κατηγορία που δημιουργεί η εισηγήτρια. Δεδομένα που δεν απαιτούν διαδικασία κοινοποίηση, δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται σε ένα σχέδιο κειμένου, ένα σχέδιο ηλεκτρονικού μηνύματος που δεν έχει καν αποσταλεί. Αυτό είναι ένα τρόπο επικοινωνία των ε, εγκληματιών, αλλά δεν εντάσσονται στην πρόταση της εισηγήτρια. Μετά, το ένταλμα παράδοση δεδομένων. Ένταλμα παραγωγής ή ένταλμα ε, διαφύλαξης στοιχείων. Πρέπει να έχουμε διάκριση μεταξύ αυτών ανάλογα με το επίπεδο της παρέμβασης. Δεν είναι τα ίδια αυτά. Όταν μιλάμε για την προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων και στοιχείων, ε, η συγγήτρια αναφέρεται στην εκτελεστική αρχή, η οποία εκτελεστική αρχή αρνείται να εφαρμόσει το ένταλμα διαφύλαξη στοιχείων. Το καταλαβαίνω, είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Ναι αλλά μία αναγνώριση ή μία άρνηση εντάλματος διαφύλαξη στοιχείων. Αναφέρεται ότι αυτή η διαφύλαξη των στοιχείων πρέπει να είναι αυτόματη. Εγώ θα προτιμούσα να δω κάτι άλλο. Να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει προθεσμία 60 ημερών που θα μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία των 60 ημερών ή να αγνοείται πλήρως, να καταργείται. Αυτή η περίοδος η χρονική των 60 ημερών που αναφέρατε θα πρέπει να είναι περιορισμένη, να μπορεί να περιοριστεί αν υπάρχει ένταλμα παραγωγής στοιχείων όπου εκτελεστική αρχή δεν είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη σχετικότητα που έχουν τα στοιχεία με μια διεξαγόμενη έρευνα. Θα πρέπει να καταβάλλεται μία προσπάθεια όμως αποφυγής απώλειας των στοιχείων. Η συγγήτρια θα ήθελε η εκτελεστική αρχή να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση εντάλματος όποτε αυτή η άρνηση εδράζεται επί συγκεκριμένων λόγων. Είναι δικαιολογημένη, είναι τεκμηριωμένη. Αυτό πρέπει να συνάδει με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Αλλά το άρθρο 10α που προσθέτει η εισηγήτρια δεν αντιστοιχεί στις ιδιαιτερότητες του είδους των στοιχείων που συζητούμε. Μιλάμε για ένα κατάλογο λόγων για μη εκτέλεση ενός εντάλματος, άρνηση εκτέλεσης ενός εντάλματος. Η συγγήτρια λέει ότι η προτινόμενη οδηγία πρέπει να απορριφθεί και θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στους νομικούς εκπροσώπους. Είναι περιπλοκότατο αυτό το εργαλείο, το αναγνωρίζω. υπάρχει μενία στους νομικούς εκπροσώπους στον κανονισμό. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίζει νομικό εκπρόσωπο του παρόχου υπηρεσιών, να αναγνωρίζει νομικούς εκπροσώπους του παρόχου που θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να συμμορφώνονται με τις αποφάσει με τα εντάλματα αν ο νομικός εκπρόσωπος είναι υπεύθυνο για παραλαβή αυτών και χρήση αυτών. Καλύτερα αυτοί οι νομικοί εκπρόσωποι παρά ο ίδιος ο πάροχος υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να το δούμε ενδελεχέστερα. Κλείνω ότι το διπλό αξιόπινο αν πρόκειται να αφαιρεθεί ε, δυσκεραίνεται ο έλεγχος, ο συνταγματικός και ο νομικός. Αν επιβάλλουμε κυρώσεις, ποινές, όταν ένα ευρωπαϊκό ένταλμα παραγωγής και διαφύλαξης στοιχείων χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα. Αν το αδίκημα στο εκδίδον κράτος, που έχει διαπραχθεί στο εκδίδον κράτος, δεν θεωρείται ποινικό αδίκημα στο κράτος που εκτελεί, αυτό θα είναι τελείως καινοφανές αν συμβεί. Δεν θα έχει παράλληλο σε άλλα εργαλεία αμοιβές αναγνώριση. Πρέπει προσεκτικότατα να εξετάσουμε τη θέση που θα ε, τηρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, τονίζω ότι συνεργαστούμε επικοδομητικά Θέλουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά με την εισηγήτρια για να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο έγγραφο, το οποίο είναι κάτι που απαιτείται, που χρειάζεται, το καταλαβαίνω. Από την αριστερά και από τη δεξιά θα καταβάλουμε προσπάθειες για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά για την επίτευξη των λόγων στόχων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ βλέπουμε ότι νομικές πράξεις που έχει ε, εκπονήσει η Κομισιόν, δυο νομοθετικές πράξεις μάλιστα εδώ που συνδέονται μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά πολιτικά, τεχνικά και νομικά προβλήματα ε, Βεβαίω και η συγκίτρια κυρία Ζίπελ και ο κύριος Μπέλο ε, χρειάστηκαν 15 λεπτά ο καθένας ε, για να μας πούν τις απόψεις τους. Ελπίζω να μην ισχύει το ίδιο για τους ε, σκιώδες γιατί ε, δεν θα προλάβουμε. οι διερμηνείς θα μας αφήσουν, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε κάπως πιο σύντομοι οι υπόλοιποι ομιλητές. Ο κύριος Κέρνερ ε, για τη Renew. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα πω λίγο πιο σύντομα όμως όπως είπατε είναι τόσο περίπλοκο ε, το μέσο αυτό που είναι δύσκολο να είναι κανείς σύντομος. Ε, και είναι τόσο περίπλοκο που θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Birgit, την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της. Είναι μια πολύ καλή βάση το κείμενο αυτό επί της οποίας μπορούμε να, μπορούμε να εργαστούμε για να φτάσουμε σε ένα σωστό συμβιβασμό στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Σε γενικέ γραμμέ ε, υποστηρίζω το στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όμω ε, αυτή η προσέγγιση ε, μία λύση για όλου ε, δεν ταιριάζει. Αυτό είναι ένα κορσέ για όλου θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη μεταρρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν προσπάθησε ε, να το διευρύνει κιόλα, ίσω κάπω υπερβολικά. Γιατί το χρειαζόμαστε, εν διότι σε κάποιου τομεί τα νομοθετικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα είναι πολύ απλά για να εξασφαλίσουν ότι θα έχουμε τα δεδομένα έγκαιρα για να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα. Ε, ο λόγο είναι λοιπόν ότι έχουμε την ενιαία αγορά για τις ψηφιακές εταιρείες, έχουμε ένα ψηφια, ψηφια, μια ψηφιακή αγορά, ένα ψηφιακό κόσμο, ε, διασυνοριακό εμπόριο, έχουμε όμως 28 εθνικά συστήματα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση για να λύσουμε, για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, χωρίς να δημιουργούμε όμως νέα προβλήματα και χωρί βεβαίω να διακυβεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποβολή του νόμου δεν πρέπει να ε, περιοριστεί λόγω αυτή τη ψηφιακή αγορά και δεν πρέπει οι εγκληματίε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά μα. Έτσι λοιπόν, για τις περιπτώσεις όπου ο, υπάρχει υποψία ε, εγκλήματος ε, ο εγκληματίας, ε, το δικαστήριο, ο, τρόπο, τόπος είναι το ίδιο, αλλά υπάρχει μόνο ένα στοιχείο που είναι εκτός της χώρας αυτής, ε, τότε οι αρχές που συλλέγουν τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να τα συλλέξουν όσο εύκολα τα συλλέγουν σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Επίσης νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τις επίγουσες περιπτώσεις. Είπε επίση ο κ. Μήλο κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Να αξιολογήσουμε την κατάσταση ε, να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι αυτός ο ύποπτος και όταν ο μόνος σκοπός είναι να, τον, να ταυτοποιήσουμε ποιος είναι αυτός ο ενδεχόμενος εγκληματίας, ε, ένας περιορισμένος αριθμός κατηγοριών δεδομένων πρέπει να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από σήμερα. Όμως, με αυτά τα τρία μέτρα, οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις ε, καλύπτονται. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, που είναι λίγες βέβαια, αλλά που είναι ευαίσθητες από πλευρά των δικαιωμάτων, πρέπει να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε ε, στον ε, ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή διαταγή ε, έρευνας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αποθηκεύουμε τα δεδομένα και να χρησιμοποιούμε τα συστήμα, το σύστημα αυτό, αυτή την, την, αυτό το μέσο. Και για να μην υπάρξει κατάχρηση κάποιου νέου εργαλείου ε, ε υπάρχει ένα κράτο μέλο στο οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία άρθρο 7. Έτσι, οπότε πρέπει να, να προσέχουμε ιδιαίτερα ε, ποια είναι η χώρα που θα κάνει αυτή την εφαρμογή πριν χορηγηθούν τα δεδομένα αυτά. Το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό το θέμα του κράτου δικαίου και ε, υπάρχουν εδώ ζητήματα θεμελιών δικαιωμάτων Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το κράτο δικαίου θα εφαρμόζεται και θα ισχύει και στις χώρες αυτές όπου ε, λαμβάνουν χώρα αυτές τις σημαντικές αλλαγές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν αλλαγές, μπορούμε να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση, να φτάσουμε σε ένα σημείο ισορροπίας. Επίσης πιστεύω ότι κάποιες από τις αλλαγές ε, που έχει επιφέρει η συγκήτρια, ε, παραδείγματος χάρη τα κατόφλια, το χρονικό όριο, οι πληροφορίες για το χρήστη, τα ένδικα μέσα, όλα αυτά τα υποστηρίζουμε. Όμως κάποιες από τις αλλαγές αυτές, ε, για κάποιες αλλαγές αυτές πρέπει να βρεθεί στο σημείο ισορροπίας, να αντιμετωπίσουν, να, να την κλιματικότητα, να προφυλάξουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ευρωπαϊκές εταιρείε, την ενιαία αγορά. Ε, πιο σημαντικό όμως είναι να εξασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους. Και πραγματικά περιμένουμε με την μονησία τη συνεργασία μα. Πιστεύω ότι θα βρούμε σημεία σύγκληση και αναμένω να συνεργαστώ με του άλλου και του και με την εισηγητριά μα για να βρούμε ένα, φτάσουμε σε ένα εργαλείο το οποίο να είναι νομικό υγιέ, να, να πετυχαίνει το στόχο του και να σέβεται ταυτόχρονα και τη θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ταρντίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Α, συγγνώμη. Ε, Πρώτα η πράσινη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ο κ. Λακοντίνσκι, ο Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουν χρόνο συνάδελφοι από την ID να μιλήσουν μετά. IND. Θα ήθελα να είμαι σχετικά σύντομο, πολύ ότι πολλά ήδη ελέγχθησαν. Βεβαίω να ευχαριστήσουμε την συνάδελφο την κυρία Ζίπελ. Είναι γιγάντιο το έργο που έχει φέρει σε πέρα και αναμένουμε να έχουμε μια καλή διαπραγμάτευση και να προχωρήσουμε. Εμείς υποστηρίζουμε τη θέση σας για τις διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά το cloud ε, στην συνθήκη με τους Αμερικανούς και με άλλες χώρες. Ε, καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει εάν δεν ολοκληρώσουμε εμείς τη θέση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ θα πρέπει να διαπραγματευτούμε πρώτα αυτή τη θέση της Ευρώπης. Και ελπίζω η Κομισιόν πραγματικά να ακούσει εδώ την εισηγήτρια και να το λάβει υπόψη της. Ε, συμφωνούμε επίσης ότι αφορά την ξεχωριστή οδηγία για την νομική εκπροσώπηση. Δεν βλέπουμε γιατί αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστού εγγράφου. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα μαζί σας. Ε, υπάρχουν μια σειρά από σημεία τα οποία πάνε προς σωστή κατεύθυνση κατά την απόψή μας. Ε, υποστηρίζουμε να υπάρχει ένας ορισμός των δεδομένων που να συνάδει με προηγούμενα κείμενα αλλά και με τις προδιαγραφές που προβλέπονται, τα πρότυπα που προβλέπουμε εμείς εδώ, οι υπάρχουσες προτάσεις απέκλειναν από αυτά και κάναμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή κατεύθυνση με αυτήν την πρόταση της εισηγήτριας. Η προστασία όσων πλήττονται ε, θα πρέπει να είναι η οχρογωνίας λίθος του σχεδίου μας. Ε, όχι μόνο η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Υποστηρίζουμε επίσης ε, την πρότασή σας ε, να μην φορτώσουμε υπερβολικά τους παρόχους με νομικές διαδικασίες. Θα πρέπει να βρεθεί ένα σωστό, σωστό σημείο ισορροπίας. Υπάρχουν κρατικές αρχές που μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα κάποιες ε, βεβαίως ε, ακραίες περιπτώσεις ε, παρανομίας και διακρίσεων θα πρέπει ήδη ο πάροχος να το εντοπίζει και να το φιλτράρει. Αυτό που λείπει όμως είναι μια εφαρμογή των αρχών της χώρας υποδοχής στο pre-screening. Βεβαίω ξέρω ότι κάνετε μια πρόταση ισορροπημένη, προσπαθείτε να βρείτε ένα συμβασμό μεταξύ των θεμελιών δικαιωμάτων του κράτου δικαίου αφενό και τη αποτελεσματικότητα από την άλλη, αλλά δεν συμφωνούμε ότι αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει βεβαίω να συζητήσουμε πώ θα πρέπει να εκπονήσουμε μια λύση που είτε θα πηγαίνει ε, προς ε, μια λύση quick trees είτε θα δίνει στη χώρα υποδοχή και σχετική αρχή το δικαίωμα και την υποχρέωση να πάρει θέση για το θέμα. Όχι να τους δίνουμε απλά χρόνο να πούν κάτι, να μην πούν τίποτα, διότι εκεί υπάρχει κίνδυνος οι περισσότερες αρχές να μην πούν απολύτως τίποτα. Ε, και ουσιαστικά ε, πάμε πίσω εκεί που θέλει να πάμε το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Ε, ή να πρέπει να βρούμε μια πολυμερή λύση για μια αρχή που θα αναλάβει αυτό το καθήκον. Πολλά λοιπόν είναι τα θέματα προς συζήτηση. Ε, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο άχθος. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και την κοινωνία των πολιτών, τις μικρές οργανώσεις, ε, τους μικρούς παρόχους, όχι μόνο τους μεγάλους που είναι στην Ιρλανδία. Ε, δεν είναι αυτό το μοντέλο μας. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε κατά νου δηλαδή και τους υπόλοιπους. Οπότε ναι, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, σημαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά, όμως αυτό που δεν θέλουμε είναι να έχουμε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ε, σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εκεί συμφωνώ και με τον κύριο και τον προηγούμενο μιλτή και τον σχέδιο τον κύριο Κέρνερ, ότι αυτό θα είναι το βασικό σημείο που θα μα απασχολήσει, αυτό θα είναι το σημείο αφετηρία μας. Αναμένω λοιπόν τι διαπραγματεύσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία. Έως τώρα έχει γίνει μια καλή αρχή, προ τη σωστή κατεύθυνση και είμαι αισιόδοξο. Σύντομα θα βρούμε αυτό το σημείο ισορροπία που θα μπορούμε να δεχτούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχετε το λόγο κυρία Ταρντίνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πάω Κατευθείαν σε ευχαριστίες προς τη συνάδελφο. Έκανε τεράστια δουλειά. Είναι θεμελιώδες ζήτημα. Πολύ σημαντικό. Πάω στα θέματα που πιστεύουμε πιο ασαφή προς διευκρίνηση. Κοινοποίηση. Συστήθηκε εκτενώς η κοινοποίηση. Στο αρχικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπεται κοινοποίηση στην αρχή του άλλου κράτου μέλους, στη στιγμή της έκδοση του εντάλματος. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν επέκταση του μηχανισμού κοινοποίηση των εντάλματων προ την αρχή του κράτου εκτέλεση. Με διαφορετικό τρόπο. Πιστεύουμε ότι η γνώση του εντάλματο από πλευρά του κράτου που εμπλέκεται θα είναι κάτι σκόπιμο για να επιτρέψει την έγκριση άρση κάποιων εμποδίων που δεν γνωρίζει η χώρα έκδοσης του εντάλματος. Πιθανότατα οι δέκα ημέρες που αναφέρονται από τη συνάδελφο είναι υπερβολικό χρονικό διάστημα. Προτείνουμε να μειωθεί στο μισό για την κατηγορία των δεδομένων. Η συγγήτρια προτείνει τρεις εγγραφές κυκλοφορία περιεχόμενου, συνδρομητές μάλλον πρώτοι, Όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ορισμός των κατηγοριών των δεδομένων είναι ένα θέμα προ επεξεργασία για να εξαλείψουμε αμφισημίες και βεβαιότητες όσον αφορά ε, το είδος κάποιων πληροφοριών, όπως η διεύθυνση ICP. Πιστεύω ότι οι διάφορες ε, διατάξεις προβλέπουν υποχρώσεις και δικαιώματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πληροφορίες ε, αυτές που ζητούνται από την δικαστική αρχή, τα δικαιώματα των ανθρώπων των ενδιαφερομένων. Η συγγήτρια έχει διάφορες προστίκες και διευκρινήσεις που κάνει για να βρεθεί μια απάντηση για το πρόβλημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προβλέπεται επικαιροποίηση συστήματο κοινοποιήσουν σωστοί ενδιαφερόμενοι ε, να προστατεύονται σε περίπτωση ελοπής εντολή από το κράτος εκτέλεσης. Θα πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκείνου που κατέχει στοιχεία που διερευνώνται. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αίτημα. Θα πρέπει όμως οι πορισμένες συγκεκριμένε περιστάσεις να ισχύει αυτό. Ίσως η άμεση γνωστοποίηση Ίσως είναι κάτι που πρέπει να κρίνεται από τη δικαστική αρχή. Μετά τα όρια των ποινών. Ελάχιστη τριετής ε, ποινή κράτηση αυξάνεται και προβλέπεται σαν πέντε χρόνια κράτησης. Επιλογή για τα όρια των ποινών πρέπει να αποτέλεσμα συγκριτικής αξιολόγησης διαφόρων εθνικών ποινικών κώδικων. Μπορεί να γίνει χάρη στην υποστήριξη της νομικής μας υπηρεσίας αυτό. Να δούμε ποια ίδια δικήματα αποκλείονται από το πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας, της νομοθεσίας, σε περίπτωση αύξηση των ποινών από τρία έτη σε πέντε χρόνια, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται το μέσο αυτό για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων με αναλογικό τρόπο και να προστατεύονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να κάνουμε και ενδελεχέστερη ανάλυση του κειμένου και των δεχομένων συνεπιών που έχουν οι τροποποίησεις που προτείνει η συγγήτρια. Όσον αφορά την πρόταση οδηγία για να αναγνωρισμένε προδιαγραφέ για του νομικού εκπροσώπου, για του σκοπού τη απόκτηση αποδείξεων σε ποινικέ διαδικασίε, είπε η συγγήτρια ότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των δύο νομικών μέσων. Στην πρόταση αυτή Υπάρχουν μέτρα συνοδευτικά όσον αφορά την αναγνώριση. Δεν θα πρέπει το περιεχόμενο μιας οδηγία να ανέβει σε επίπεδο κανονισμού. Είναι υπερβολικό. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή τη υποχρέωση καθορισμού νομικών εκπροσώπων με άλλο τρόπο. Γιατί με αυτό που προτείνεται δημιουργούνται προβλήματα. Πιο ευέλικτη οδηγία επιτρέπει στα κάτι μέλη να χρησιμοποιήσουν την νομοθεσία μεγαλύτερη ευελιξία. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν τρόποι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, τροποποιώντας το, να δούμε ποια κράτη-μέλη δεσμεύονται από την υποχρέωση για το διορισμό νομικών εκπροσώπων. Μπορούμε να δούμε με την νομική υπηρεσία. Σε σχέση με τη θέση Δανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα νομικός πώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω σκιώδη ηγητή από την Ενωτική Αριστερά να μας παρουσιάσει την άποψη της ομάδας. Επανερχόμαστε στην εισηγήτρια. And, uh, uh, Σημειώσατε όλα τα σχόλια, κυρία Ζίπελ, σίγουρα. Και όλες τις διαπραγματευτικές ε, τακτικές. Αλλά προηγουμένως να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σίγουρα θα θέλει και αυτή να απαντήσει. Ευχαριστώ. Να μιλήσω σύντομα. Δεν θέλουμε να πούμε σε λεπτομέρειες απόψε. Ευπρόσδεκτη η έκθεση, το σχέδιο εκθέσεως. Σημαντικό να προχωρήσουμε στις συζητήσεις μας. Υπάρχουν και διεθνείς πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχουμε κάτι στα χέρια μας είναι βάση συζητήσεων. Να επενθυμίσω κάτι. Αφετηρία μας, όταν κάναμε την πρότασή μας, για τα δύο εργαλεία και το πακέτο, ήταν να ασχοληθούμε με το πρόβλημα που έχουν οι ερευνητικέ αρχές. Δεν έχουν πρόσβαση πλέον σε αυτά τα στοιχεία. Αρκετά, δεν έχουν ταχεία πρόσβαση, επαρκώς ταχεία. Και καθόλου πρόσβαση. Όταν συμβαίνει αυτό και έχουν χαθεί τα στοιχεία, τι γίνεται. Μετά τον Μπατακλάν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και σε άλλες επιθέσεις μετά. Οι άνθρωποι του κλάδου ζήτησαν από τους Ευρωπαίους νομοθέτες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν κάτι. Να τους δώσουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Να είναι πιο χρήσιμο από τα παρόντα εργαλεία. Δεν λέμε ότι η αποδοτικότητα είναι το παν. Συμφωνούμε με αυτό που είπαν πολλοί αγορητές. Χρειάζεται επαρκής προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Αν δεν πετύχουμε αποδοτικότητα με αυτό το μέσο, χάνουμε το σκοπό του μέσου, να έχουμε βελτιωμένο μέσο. Έχουμε ανησυχίες όσον αφορά τις προτάσεις του σχεδίου εκθέσεως. Η διαδικασία περιπλέκεται περαιτέρω. Πρέπει να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες. Βλέπω πολλές επιπλοκές και περιπλοκές συμπεριλαμβανομένου του συστήματος κοινοποίησεως με την εμπλοκή τριών διαφορετικών κρατών μελών, άρα εμπλέκονται τρει και ενδεχομένω τέσσερι ένομε τάξει. Και ίσω να υπάρχει και σύγκρουση με την νομοθεσία τρίτη χώρα. Υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε που αποδυναμώνουν την πρόταση. Χάνει την προστιθεμένη αξία τη. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε Για την οδηγία να πω κάτι. Γιατί προτείναμε δύο εργαλεία. Όχι θεωρήσαμε ότι δύο είναι καλύτερα από ένα, για νομικού σκοπού το κάναμε. Συμπεράναμε ότι κυρίως όσον αφορά τους παρόχους τρίτων χωρών, η νομική βάση του άρθρου 82 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή υποχρεώσεων σε αυτούς διότι δεν μιλάμε πλέον για δικαστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, μιλάμε για παρόχους τρίτων χωρών. Το άρθρο 82, βάσει της δικής μας νομικής αναλύσεως που έγινε τότε, δεν είναι η κατάλληλη νομική βάση. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα αν ενσωματώσουμε αυτές τις διατάξεις στον κανονισμό. Τούτου λεχθέντος με τα χαράς να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές για να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Αν επιθυμείτε μια συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στην εισηγήτρια. Ακούστηκαν τα σχόλια στα όσα είπατε. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε. Εγώ να πω Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Μετά. Έχετε το λόγο κύριε Συγήτρια. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. με λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσω ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχομένω και τρίτη και τέταρτη ενδεχόμενη χώρα. Τι δείχνει αυτό τελικά, ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό και δεν μπορούμε παρεπιπτόντως να αποφασίσουμε μια νέα προσέγγιση. Συμφωνώ επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση IP, δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να εμπλακεί άλλη χώρα. Αλλά εκπλήσωμε, τώρα μιλάμε για ένα νέο νομοθέτημα. Το νέο νομοθέτημα θα πρέπει να ε, είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις περιπτώσεις. Πολύ συχνά μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άκουσα και σκιώδης να λένε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ε, ε, το έγκλημα γίνονται στη χώρα που εκδίδει και την εντολή και εκεί διαμένουν και οι ε, ύποπτοι. Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου το έγκλημα δεν διαπράτεται τελείως στην εκδίδουσα χώρα, ούτε διαμένει ε, ο υπόπτος εκεί. Θα πρέπει να λειτουργεί αυτό το εργαλείο σε όλες τις περιπτώσεις και να μην ε, παραλείπτει κάποια πράγματα. Ε, θα, έχω να πω και άλλα, αλλά δεν θα το κάνω σήμερα. Θα το συζητήσω με τους κοιόδης μας συγητές και θα το βρούμε. για το χρονοδιάγραμμα νομίζω μάλλον τις προθεσμίες δεν τα αυξήσαμε. Κάποιος συνάδελφος είπε ότι 10 ημέρες είναι υπερβολική προθεσμία. Μα αυτό προτείνει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Εμείς δεν παρατείνουμε εκεί αυτή την προθεσμία. Σε ό,τι αφορά το θέμα τώρα, αν θα είναι οδηγία ή κανονισμός, regulation, έχει περάσει η κανονισμος regulation εχει περασει ωρα δεν θυμάμαι και στα αγγλικά πώς λέγεται ο κανονισμός. Αν θέλουμε όμως να εναρμονίσουμε τους κανόνες και να έχουμε ένα νομικό μέσο που να ε, προσφέρεται για όλες τις περιπτώσεις και να το ακολουθούν όλοι, δεν μπορούμε από την άλλη να έχουμε οδηγία που είναι στον πατριωτισμό των κρατών μελών, αν θα το εφαρμόσουν και πώς. Ε, γι' αυτό είναι επιπλέον λόγος να γίνει ε, ε, κανονισμός και όχι οδηγία και να συμπεριληφθεί εκεί. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία των δεδομένων, πολύ ενδιαφέρουσα αναμένεται η ανταλλαγή απόψεων, καθώς επίσης και ο ορισμός. Τη διαφορά ε, υπάρχει όταν μιλούμε για δεδομένα σχέση με το περιεχόμενο, αν έχουν ήδη αποσταλεί, αν είναι ακόμα στο σερβερ. Γιατί το περιεχόμενο έχει δύο διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων ανάλογα με το που βρίσκεται. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να κανονίσουμε ε, συνεδριάσεις οδών που να μπορούν να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι για να ανταλλάξουμε απόψεις για τα θέματα αυτά που ακούσαμε σήμερα και ενδεχομένως και κάποια άλλα που δεν αναφέρθηκαν. Για να δούμε τώρα πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Α, ένα συμπληρωματικό. Δεν άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόλου να μας λέει αν διαπραγματεύονται σε λεπτομέρειες με τις Ηνωμένε Πολιτείε για το θέμα αυτό με βάση τη δική τους πρόταση προεξοφλώντας ενδεχομένως την απόφαση που θα πάρουμε εμείς για τα ηλεκτρονικά αποδεκτικά στοιχεία. Έχει να απαντήσει τίποτα σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, δεν προδικάζουμε τίποτα στις αρχικές μας συζητήσεις με τους Αμερικανούς. και είναι διαφορετική και η κατάσταση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί αναφέρονται συνέχεια διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Οι συζητήσεις εκεί θα χρειαστούν πολύ χρόνο. Έχουμε δεσμευτεί, νομίζω, να μην ολοκληρωθεί τίποτα πριν διαθετηθούν οι εσωτερικοί μας κανόνες. Και γνωρίζουμε ότι είναι η βάση μας οι εσωτερικοί κανόνες. Και αυτή είναι η εντολή μας. βασιζόμαστε στου εσωτερικού κανόνε όπω αυτοί εξελίσσονται στη θητεία μα για τι διαπραγματεύσει. Στι διαπραγματεύσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη δεν προδικάζουμε τίποτα. Ούτε εμεί θα καθορίσουμε όμω το ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ενό έτου πριν εκπνεύσουν οι προδιαγραφέ τη εντολή τη διαπραγματευτικής ομάδα. Έχουμε ένα χρονικό όριο που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε βάσει των εσωτερικών μας κανόνων που είναι η αποκλειστική μας βάση για τις διαπραγματεύσεις και για τυχόν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο. Αρκεί, φτάνει για τώρα. Λοιπόν, μόλις συζητήσαμε το σχέδιο έκθεσης και μόνο που κατέθεσε η συγγήτρια. Κάναμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις. Το μόνο που μπορούμε τώρα να κάνουμε είναι να ορίσουμε μια προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών 27 ενδεκάτου, 5 η ώρα το απόγευμα. Η έγκριση του σχεδίου έκθεσης και η ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης στην Ολομέλεια δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Μόνο η προθεσμία για τις τροπολογίες 27 ενδεκάτου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 για τη συνέχεια. Και σας θυμίζω ότι το πρωί έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ να φέρετε τις κάρτες σας. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.